Παρακαλώ, κάντε λίγη ησυχία για να μπορέσουμε να αρχίσουμε την απογευματινή μας ε, συνεδρίαση. Όπως σα ε, σας είχα πει το πρωί, έχουμε τη χαρά να καλωσορίσουμε στη συνεδρίασή μας τον Υπουργό Αθανάσιο Τσαφτάρη Υπουργό της Αγροτικής Ανάπτυξης, Υπουργό της Ελληνικής Κυβέρνησης. Όσοι ήθιστε, σας υποδεχόμαστε στην Επιτροπή μας στις απαρχές της Προεδρίας. Με μεγάλη χαρά θα σας ακούσουμε. Δεν θέλω να χάσουμε χρόνο. Μόνο να σας πω ότι έχουμε μία αντιπροσωπεία γεωργών από την Πορτογαλία που παρακολουθούν τη συνεδρίασή μας εδώ μέσα στην αίθουσα. Καλώς ορίσατε κι εσείς. Η κυρία Πατραονέβες έχει προσκαλέσει την ομάδα των επισκεπτών. Και μετά τη μεταρρύθμιση της κοινή ε, γεωργικής ε, πολιτικής κατά την περίοδο εφαρμόγης ε, θα υπάρξουν και άλλες τέτοιες επισκέψεις. Δίχως περαιτέρω καθυστέρηση, θα ήθελα να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι ε, τα μέλη της Επιτροπής μας ενδιαφέρονται πάρα πολύ για οποιασδήποτε πληροφορίες μπορείτε να δώσετε για το πρόγραμμα της ελληνικής κυβέρνησης στον τομέα της γεωργίας, κυρίως ως προς την εφαρμογή ακριβώς ε, της κοινής γεωργικής πολιτικής ε, που μεταρρυθμίσαμε πρόσφατα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει σε αυτό το τομέα. Εργάστηκε επί σειρά μηνών για να καταθέσει τροπολογίες στο σχέδιο μεταρρύθμισης κοινής γεωργικής πολιτικής. Εξάλλου πολλές αλλαγές ε, πηγάζουν από τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα έχουμε εισέλθει στην περίοδο εφαρμογής της μεταρρυθμισμένης κοινή γεωργικής πολιτικής και πλέον τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν αναλάβει την εφαρμογή αυτής της νέας πολιτικής. Φυσικά πολλά θα εξαρτηθούν από την τρέχουσα ελληνική προεδρία. Σας δίνω τον λόγο ευθύ αμέσως. Παρακαλώ. Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι και αγαπητοί αγρότες. Είναι για μένα μεγάλη τιμή που βρίσκομαι εδώ σήμερα με την ευκαιρία της ανάληψης της πέμπτης ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να παρουσιάσω το πρόγραμμά μας στην Επιτροπή Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να συζητήσουμε με τον νομοθέτη του Συμβουλίου που διαθέτει πλέον μεγαλύτερη επιρροή προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας και φυσικά προς όφελος των Ευρωπαίων αγροτών. Μιλώντας για την γεωργία και την αλληλεία, μιλούμε για το τον πρωτογενή πλούτο της Ευρώπης. Έναν πυλώνα ανάπτυξης και απασχόλησης, ένα τομέα που εξασφαλίζει την εξαιρετική ποιότητα της διατροφής μας με σεβασμό στους φυσικούς πόρους και στην κοινωνία. Επιτρέψτε μου να αναφέρω πρώτα συνοπτικά τις οριζόντιες προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας. Πρώτον, η τόνωση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της συνοχής. Το ένα προϋπόθεση του άλλου που μπορούν να συμβαδίσουν αρμονικά με την δημοσιονομική πειθαρχία. Δεύτερον, τη στήριξη του νομ... κοινού νομίσματος και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης της κοινωνίας και των πολιτών στην ευρωπαϊκή ιδέα. Τρίτον, οι εξωτερικές προκλήσεις και η απάντηση που οφείλει να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μεταναστευτικό ζήτημα, η τραγική διάσταση του οποίου αναδεικνύεται συχνά στη θαλάσσια, στα θαλάσσια και τα χερσαία σύνορα της Ευρώπης. Τέλος, η ελληνική προεδρία φιλοδοξεί να δώσει νέα πνοή στις θαλάσσιες πολιτικές της Ένωσης. Μια θεματική που διατρέχει βέβαια οριζόντια τις προτεραιότητές μας. Ερχόμενος τώρα στη Γεωργία, αναλαμβάνουμε την Προεδρία σε μια περίοδο μεταβατική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την κοινή αγροτική πολιτική. Εγκρίναμε, όπως τόνισε και ο κύριος Πρόεδρος, πρόσφατα τη μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής και πρέπει τώρα να φροντίσουμε η μετάβαση στη νέα κατάσταση να είναι ομαλή και να διευκολύνει τους γεωργούς στην παραγωγική τους δραστηριότητα και φυσικά στις επενδύσεις τους. Ταυτόχρονα πρέπει να αξιολογήσουμε ορισμένα μέτρα της κοινή αγροτικής πολιτικής και να εντοπίσουμε τις αναγκαίες βελτιώσεις, να ενισχύσουμε τη θέση των αγροτών και των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων στην εμπορική διαδικασία. Να τους φέρουμε πιο κοντά στον καταναλωτή. Είναι αναγκαίο να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα και κάθε εργαλείο που πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει ώστε η γεωργία να είναι αποδοτική για τους γεωργούς, φιλική για το περιβάλλον και την κοινωνία και αξιόπιστη για τους καταναλωτές. Η ποικιλομορφία αποτελεί γνώρισμα και συγκριτικό πλεονέκτημα της ευρωπαϊκής γεωργίας και της χώρας μου και πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Τα ποιοτικά αναγνωρίσιμα πιστοποιημένα και ασφαλή προϊόντα που αντανακλούν τα αυστηρά πρότυπα παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ιδιαίτερη φροντίδα της οικογενειακής εκμεταλλεύσεως. Χρειάζονται μια ιδιαίτερη προσοχή. Σε αυτό το πλαίσιο διαμορφώνεται το πρόγραμμά μας. Πρώτον, πρώτο μας μέλημα, η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, της κοινή αγροτικής πολιτικής, μια μεταρρύθμιση που αποτέλεσε κοινή μας επιτυχία και τονίστηκε ήδη. Ένα εγχείρημα που κατέδειξε ότι μαζί μπορούμε να εργαστούμε αποτελεσματικά για την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Τώρα πρέπει να εγκριθούν έγκαιρα από την Επιτροπή ή κατεξουσιοδότηση πράξης όπως προβλέπονται από τη μεταρρύθμιση που συμφωνήσαμε. Υιοθετώντα τη μεταρρύθμιση αυτή επιδείξαμε τα τρία θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλληλοκατανόηση και πνεύμα καλής συνεργασίας. Η κατεξουσιοδοτηση πραξης οπως προβλεπονται απο τη μεταρρυθμιση που συμφωνησαμε Υιοθετώντας τη μεταρρυθμιση αυτη επιδειξαμε τα από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο που προβλέπεται από τη συνθήκη της Λισαβόνας είναι ευκαιρία για να διασφαλίσουμε ότι οι πράξεις αυτές είναι πιστές στις πολιτικές μας αποφάσεις. Η Προεδρία ευελπιστεί ότι παρά τις αρχικές ανησυχίες η Επιτροπή αφουγκράστηκε τους ειδικού των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι θα καταλήξει σε κατεξουσιοδότηση πράξεις που αντανακλούν πιστά την πολιτική μας συμφωνία σχετικά με τους νέους κανονισμούς της κοινή αγροτικής πολιτικής. Έτσι, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να είμαστε σε θέση να συμφωνήσουμε παρέχοντας με τον τρόπο αυτό στους γεωργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα σταθερό περιβάλλον. Ο φάκελος της προώθησης των αγροτικών προϊόντων είναι επίσης προτεραιότητα για την ελληνική προεδρία η συζήτηση στο Συμβούλιο είναι σε πρώιμο στάδιο. Καλωσορίζουμε την πρόταση της Επιτροπής που επιχειρεί να εξυγχρονίσει και να ενισχύσει το καθεστώς της προώθησης και είμαστε σίγουροι ότι μαζί τα τρία θεσμικά όργανα μπορούμε να βρούμε τις καλύτερες λύσεις για τους παραγωγούς αλλά και τους καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κόσμου. Μια και το πρόγραμμα αφορά και την εξωστρέφεια των ευρωπαϊκών προϊόντων. Είμαστε ρεαλιστικοί στις φιλοδοξίες μας και πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε προσεκτικά προκειμένου να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Προτείνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εργαστούμε παράλληλα ανταλλάσσοντας και τακτικά πληροφορίες ώστε να έχουμε την μέγιστη δυνατή πρόοδο και να έχουμε μια ισχυρή βάση και ίσως κατάληξη των διαπραγματεύσεων κατά το δεύτερο εξάμενο του 2014. Ο τομέας των φρούτων και λαχανικών είναι σημαντικός για πολλές περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την οικονομία της και για την υγιεινή διατροφή. Στο Συμβούλιο σκοπεύουμε να εξετάσουμε προσεκτικά την έκθεση που αναμένουμε από την Επιτροπή το πρώτο τρίμηνο του 2014 για τα αποτελέσματα της αναθεώρησης του 2007 και να καταλήξουμε σε χρήσιμα συμπεράσματα για το μέλλον αυτού του τόσο σημαντικού τομέα. Ο γαλακτοκομικός τομέας είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικός για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την οικονομία αλλά και την απασχόληση. Η Ελληνική Προεδρία έχει ήδη απαντήσει θετικά στην πρόσκληση της Επιτροπής να συζητήσει στο Συμβούλιο το πρώτο τρίμηνο του 2014 σχετικά με το μέλλον του τομέα και τον Ιούνιο του 2014 σχετικά με τα αποτελέσματα της εφαρμογής του γαλακτοκομικού πακέτου. Οι σημερινές συνθήκες της αγοράς των γαλακτοκομικών προϊόντων είναι βίωνες και είναι ίσως η κατάλληλη στιγμή για να εξετάσουμε αν όλα τα μέτρα που έχουν υιοθετηθεί στο πακέτο του γάλακτος και στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ είναι επαρκή σε περιπτώσεις κρίσης και ιδιαίτερα όσον αφορά τις μειονεκτούσες περιοχές όπου οι συνθήκες για την παραγωγή είναι δυσχερέστερες. Γνωρίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναλάβει ανάλογες πρωτοβουλίες όπως εκείνες για το μέλλον του τομέα των κυπευτικών και για τη διατήρηση της παραγωγής γάλακτος ιδιαίτερα όπως τονίστηκε στις ευαίσθητες περιοχές. Πρωτοβουλίες που δείχνουν πως μοιραζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες για την Ευρωπαϊκή Γεωργία. Το Συμβούλιο αναμένει σύντομα και την πρόταση της Επιτροπής για τα σχολικά προγράμματα διανομής γεωργικών προϊόντων στους μαθητές στόχος της ελληνικής προεδρίας είναι να εξεταστεί η πρόταση αυτή σε τεχνικό επίπεδο και να υποβληθεί στο Συμβούλιο η έκθεση προόδου των εργασιών μας τα αποτελέσματα της δημόσιας δηλαβούλευσης που έγινε στις αρχές του 2013 έδειξαν επίσης το ενδιαφέρον της κοινωνίας για την βιολογική γεωργία και τα βιολογικά προϊόντα της. Πολλά κράτη-μέλη είναι υπέρ της απλοποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας και η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι υπάρχουν αδυναμίες στο καθεστώς που πρέπει να επανεξεταστούν. Η Ελληνική Προεδρία λοιπόν καλωσορίζει αυτή την πρόθεση της Επιτροπής να παρουσιάσει την νομοθετική της πρόταση το Μάρτιο και είναι έτοιμη αμέσως να ασχοληθεί με τη νέα αυτή πρόταση. Η έκθεση της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός νέου προαιρετικού σήματος προϊόν νησιωτικής γεωργίας αναφέρεται στα ωφέλη και στις δυσκολίες παράλληλα που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν από μια τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία. Συμπεραίνοντας ότι οι περισσότερες δυσκολίες που, θα αντιμετωπίζουν τα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο γεωργικός τους τομέας πρέπει να αντιμετωπιστούν κυρίως από τα εφιστάμενα διαρθρωτικά εργαλεία. Θα συνεργαστούμε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με στόχο να εξετάσουμε εάν αυτή η έκθεση πρέπει να συνοδεύεται από μια κατάλληλη νομοθετική πρόταση στο Συμβούλιο θα συζητήσουμε την έκθεση αυτήν καταρχήν σε μια επόμενη ειδική επιτροπή γεωργίας. Η ποικιλομορφία της ευρωπαϊκής γεωργίας, τα τοπικά χαρακτηριστικά της ταιριάζουν στο μοντέλο των οικογενειακών εκμεταλλεύσεων που επικρατούν στις περιφέρειές της και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σημαντικές πρωτοβουλίες της κόμμα προς αυτή την κατεύθυνση όπως για τα περιφερειακά σήματα ποιότητας, και για τον μέλλον των μικρών εκμεταλλεύσεων. Το Συμβούλιο υποδέχθηκε με ικανοποίηση το πακέτο για τα ασφαλέστερα ζώα και φυτά και ασφαλέστερη αγροδιατροφική αλυσίδα που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή προκειμένου να αντιμετωπιστούν πολύπλοκα θέματα στους επιμέρους τομείς αλλά και την προσπάθεια που έγινε για τον εξυγχρονισμό του νομικού πλαισίου. Οι συζητήσεις της ομάδας εργασίας έχουν ήδη ξεκινήσει από τον Ιούνιο και η εξέταση αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη. Η ελληνική προεδρία σκοπεύει να ολοκληρώσει την τεχνική εξέταση των επιμέρους προτάσεων και να συνταχθούν τα πρώτα συμβιβαστικά κείμενα, τα οποία θα ενσωματώνουν τις απόψεις που εκφράζονται ήδη από τα κράτη-μέλη. Παράλληλα, η ελληνική προεδρία σκοπεύει να παρακολουθεί στενά το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να διευκολύνει κατά το δυνατόν τις, διοργανω... τις διοργανωτικές διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια της επόμενης κοινοβουλευτικής περίοδου. Ειδικότερα όσον αφορά την πρόταση για τον φυτικό αναπαραγωγικό υλικό, η Ελληνική Προεδρία θα εργαστεί από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επιχειρώντας να ανοίξει το δρόμο για την ανάπτυξη, επίτευξη μιας μελλοντικής συμφωνίας στον τομέα αυτό. Γνωρίζουμε πολύ καλά τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από ορισμένου βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και των πολιτικών ομάδων σχετικά με τις διάφορες προκλήσεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση. Το Συμβούλιο εξετάζει προσεκτικά την πρόταση αναφορικά με τις επιπτώσεις και τις συνέπειές της οι εκτιμήσεις αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για μια τέτοια πρόταση που έχει στόχο να εξυγχρονίσει αλλά και να απλουστεύσει ένα μεγάλο αριθμό λεπτομερών και τεχνικών μέτρων που ισχύουν εδώ και πολλά χρόνια. Βέβαια απαιτείται αρκετή προσπάθεια ακόμη ώστε να πετύχουμε σαφείς κανόνες και νομική ασφάλεια ακόμα και στη συνέχεια στο πλαίσιο των εξουσιοδιωτικών και εκτελεστικών πράξεων. Όσο αφορά την πρόταση κανονισμού για τη διαχείριση των δαπανών στον κτηνιατρικό και υγειονομικό τομέα, τόσο το Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο εργάστηκαν σκληρά για να εξασφαλιστεί η έγκρισή της πριν από το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περίοδου και για την επιτυχία της συμφωνίας σε πολιτικό επίπεδο. Η έκθεση της Επιτροπής για την υποχρεωτική αναγραφή της καταγωγής ή του τόπου προέλευσης του κρέατος που χρησιμοποιείται ως συστατικό σε τρόφιμα περιλαμβάνεται στο πρόγραμμά μας. Αναφορικά με άλλες προτάσεις που εκκρεμούν ή που αναμένονται η υποβολή τους, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε εφόσον συντρέχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη πρόοδος. Αναμένονται ακόμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι προτάσεις στους τομείς των κτηνιατρικών, φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακούχων ζωοτροφών της δέσμης για την υγιεινή και, νομοθε... και της νομοθεσίας για τα ζωοτεχνικά ζητήματα κλπ. Η ελληνική προεδρία είναι έτοιμη και εδώ να προχωρήσει στην τεχνική εξέταση εφόσον διαβεβαστούν έγκαιρα από την Επιτροπή. Όπως επίσης η Επιτροπή, η Προεδρία είναι έτοιμη να αρχίσει την εξέταση των προτάσεων σχετικά με την κλωνοποίηση των ζώων στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου. Όλοι οι φορείς που έχουν ήδη εμπλακεί στη συζήτηση γνωρίζουν πόσο ευαίσθητο είναι αυτό το θέμα. Η Ελληνική Προεδρία γνωρίζει επίσης την πρόσφατη σχετική συζήτηση στην ΚΟΜΕΝΒΗ και θα συνεχίσει να παρακολουθεί συστηματικά τις εργασίες του Κοινοβουλίου. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, αξιότιμα κυρίες και κύριοι, έκανα μια μικρή ανασκόπηση των προτεραιοτήτων της ελληνικής προεδρίας στο πεδίο των εργασιών του Συμβουλίου Γεωργίας σε μια σειρά από σημαντικά θέματα που έχουμε να χειριστούμε στους επόμενους μήνες. Στη συγκυρία των ευρωεκλογών, μια διαδικασία ιερή και δηλωτική της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που διέπει τη λειτουργία της αποτελεί για μας πρόκληση να εργαστούμε με ρεαλισμό και με την πεποίθηση για ένα καλό αποτέλεσμα. Βασιζόμαστε για το σκοπό αυτό στη στενή, την ενεργό και αποτελεσματική συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι απαραίτητη ώστε να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τους στόχους μας και να μπορέσουμε από κοινού να βρούμε λύσεις σε μια σειρά από σημαντικά και ευαίσθητα ζητήματα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Κύριε Πρόεδρε, με πολύ χαρά θα δεχτώ ερωτήσεις που ενδεχόμενα έχετε εσείς και τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ και πάλι για την προσοχή σας. Ευχαριστώ Υπουργέ για την ε, παρουσίασή σας. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα για αυτήν την ε, περίοδο της ε, ελληνικής ε, προεδρίας και του τέλους της τωρινής θητείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όλα αυτά παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίως στο πλαίσιο της μεταρρυθμισμένης κοινή γεωργικής πολιτικής. Για όλους αυτούς τους λόγους πραγματικά υπολογίζουμε στις πρωτοβουλίες και στις εργασίες του Συμβουλίου. Θα ακούσουμε πρώτα απ' όλα τους συντονιστές, ο κύριος Ντες πρώτος από όλους. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε κύριε Προεδρεύοντα, κύριε Υπουργέ, κύριε Τσεφτάρη για την παρουσία σας. και για την παρουσία των προτεραιοτήτων της ελληνικής ε, προεδρίας. Θα πρέπει πράγματι να εφαρμοστεί οριστικά τους επόμενους μήνες και η μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής και εγώ όπως και άλλοι συνάδελφοι ανησυχούμε για το ότι η Κομισιόν από ό,τι φαίνεται στις ε, πράξεις ε, κατεξοδότηση αποκλίνει από την πολιτική συμφωνία. Παραδείγματο χάρη το θέμα ενεργή γεωργή. Εάν δούμε την πρόταση της ε, Κομισιόν υπάρχει πάρα πολύ γραφειοκρατία όταν είναι να εξεταστεί παραδείγματο χάρη το ποσοστό του εισοδήματο που προέρχεται από τη γεωργία σε σχέση με άλλες πηγές. Μόνο ένα παράδειγμα θα σας φέρω από την ε, Βαβαρία. Εάν έχει κάποιος ε, ένα χωράφι 5 εκταρίων και έχει, το οποίο καλλιεργεί και μετά έχει και μία άλλη σύνταξη, ένα άλλο εισόδημα, βλέπουμε πως ε, θα του κοπεί η επιδότηση και τελικά τι θα κάνουμε, θα τιμωρήσουμε αυτούς οι οποίοι καλλιεργούν υπό δύσκολες ε, συνθήκες. Πρέπει λοιπόν νομίζω να εξεταστεί αυτό το ζήτημα, δεν νομίζω να μπορέσουμε να το επιτρέψουμε. Δεν ήταν αυτό το αντικείμενο της πολιτικής ε, συμφωνίας. Θα πρέπει να μπορούν να αποφασίζουν τα κράτη-μέλη ποιες εκτάσεις θα επιδοτηθούν και ποιες όχι. Δεύτερον, οι νέοι αγρότες αναφέρθηκαν ήδη και εδώ πέρα έχουμε ένα πρόβλημα. Στη χώρα μας ε, συχνά υπάρχουν κάποιες έτσι μικρές ή ατομικές επιχειρήσεις, ε, ένας πατέρας και ένας γιος ε, και δύσκολα αναγνωρίζονται και νομίζω και αυτά είναι στο πνεύμα της συμφωνίας. Τέλος, το λεγόμενο πρασίνισμα δεν είναι δυνατόν η Κομισιόν να κάνει προτάσεις, ε, παραδείγματος χάρη για τις πολιετής ε, καλλιέργειες, να επιτρέπεται να φυτεύονται μόνο συγκεκριμένα είδη φυτών ή δέντρων. Πρέπει εδώ πέρα και τα κράτη-μέλη να μπορούν να αποφασίζουν ποια είδη φυτών ή δέντρων θα επιτρέπονται και συνολικά όσον αφορά το λεγόμενο πρασίνισμα πρέπει να γίνουν ακόμα πάρα πολλά. Οπότε το ερώτημά μου κύριε Υπουργέ, εσείς ε, η ελληνική προεδρία θα δώσετε βάρος ε, σε στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο έτσι ώστε να εφαρμοστούν οι πράξεις κατεξιοδότηση όπως αποφασίσαμε εμείς πολιτικά και όχι όπως θέλει η κυρία Χέντεγκαρτ και ο κύριος Ποτότσνικ. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Κάπλας Σάντος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ αρχίζοντας να χαιρετήσω τον Υπουργό. Είναι η χαρά μας και τιμή μας να σας υποδεχόμαστε εδώ στο Κοινοβούλιο. Καλή επιτυχία για την Ελληνική Προεδρία θα ήθελα να ευχηθώ. Ε, είστε ε, στο ύψος του καθήκοντος που σας έχουν αναθέσει. Ε, τον περασμένο Νοέμβριο είχαμε όλοι συμμετάσχει στις διοργανικές συνομιλίες και τώρα έχουμε αναλάβει ένα διαφορετικό καθήκον για μας. Δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση. Όπως είπε ο συνάδελφος Ντες, είμαστε σε εγρήγορση σε σχέση με τις κατεξουσιοδότηση πράξεις, διότι περιέχουν πολύ σημαντικές λεπτομέρειες. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτική προσεκτική ούτω ώστε στην νομοθεσία να μην χαθεί στις λεπτομέρειες το πνεύμα αυτού που καταφέραμε μετά από ατελείωτους μήνες διαπραγματεύσεων. Ε, καταλήξαμε σε μια εξισορροπημένη συμφωνία. Καταφέραμε να προωθήσουμε την θέση του Κοινοβουλίου ε, και το Μάρτι θα είναι το επόμενο ραντεβού μας. Ε, ελπίζω να αναλάβει την αντίστοιχη δράση και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. είναι πολύ μεγάλες απαιτήσει για σας, διότι στο μισό χρόνο θα πρέπει να φέρετε σε πέρας πολύ δύσκολα καθήκοντα, διότι τέλη Απριλίου θα κλείσει τις πόρτες το Κοινοβούλιο και η επόμενη αγαπημένοι συνάδελφοι στην επόμενη θητεία ήδη ε, θα αρχίσουν να συνεργάζονται με την επόμενη Προεδρία. Είναι εξαιρετικά φιλόδοξο το πρόγραμμά σα. πολύ διεξοδική η παρουσία που μα κάνατε. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειε τις προσυπογράφω ε, τι αρχέ που θέσατε. Ήθελα μόνο να θα επιστήσω την προσοχή σα σε δύο σημεία. Μπορείτε να μα εκθέσετε το όραμά σα και το όραμα του Συμβουλίου για δύο ζητήματα. Πρώτον, ακριβώ αυτέ οι πράξει κατά εξουσιοδότηση. Πώ θα τι παρακολουθήσετε. Είναι ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα τη ε, τρέχουσας ε, περίοδου. Ε, δεύτερον, ε, κάτι στο οποίο και εσείς αναφερθήκατε, το φυτοναπαραγωγικό υλικό έχει αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά μία θέση η οποία θα μπορούσε να μας οδηγήσει ε, σε ανάθεση του φακέλου στην ε, Προεδρία. Είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα, ε, ιδιαίτερα λεπτό για να το πραγματευτούμε κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής περίοδου. Πιστεύουμε ότι θα έπρεπε με μεγαλύτερη ηρεμία να αρχίσουμε να το συζητάμε με την αρχή της νέας θητείας. Ε, Γνωρίζετε τη θέση του Κοινοβουλίου. Θα θέλαμε, κύριε Υπουργέ, ή δυνατόν να μας εκθέσετε τη δική σας άποψη για αυτό το ζήτημα. Ε, πιστεύετε ότι είναι πολιτικά πρόσφορο να συνεχίσετε τη συζήτηση τέτοιας φύσεως για ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα ως προς την κοινή γνώμη ε, σε μια τέτοια αμφιλεγόμενη περίοδο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χόσλινγκ παρακαλώ τώρα έχει το λόγο. Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, σας καλωσορίζω και εξ ονόματος των Πρασίνων και εμείς βεβαίως έχουμε ερωτήσεις για την Προεδρία σας. Μια ερώτηση είναι βεβαίως ένα ζήτημα επίκαιρο στη Γερμανία η επαναδιοδότηση του γενετικά τροποποιημένου καλαμποκιού το λεγόμενο 1507 ε, τι σκοπεύετε να κάνετε δεν μιλάω διαδικαστικά μόνο για μένα το ζήτημα είναι πως η τελευταία εξέταση αυτού του είδους έλαβε χώρα το 2009 δεν ε, επαρκεί αυτό μόνο για να ξεκινήσει μια νέα διαδικασία επανεξέτασης πριν ε, προχωρήσουμε σε επαναδιοδότηση ενός γενετικά τροποποιημένου είδους ε, καλαμποκιού και ειδικά πριν τις εκλογές. Επίσης γνωρίζετε πως η Κομισιόν ανακοίνωσε Πώς θα φέρει τέλος Μαρτίου ένα νέο κανονισμό για τα βιολογικά προϊόντα. Εγώ δεν έχω αντίρρηση για επεξεργασία του κανονισμού, αλλά όταν μιλάμε για το τέλος ε, Μαρτίου δεν είναι πολύ βολική στιγμή για τους βουλευτές για να ξεκινήσει ξανά μια τέτοια συζήτηση. Τι σκοπεύετε λοιπόν να κάνετε. Νομίζω πως δεν θα έχουμε την ευκαιρία και το χρόνο να συζητήσουμε και να τοποθετηθούμε για τον κανονισμό αυτόν. Και βεβαίως οδηγεί σε ανασφάλεια τους αγρότες αυτό όταν παρουσιάζεται ένας ε, νέος ε, κανονισμός και θα μας απασχολήσει τελικά στο τέλος του έτους. Αναφερθήκατε στην κλωνοποίηση ε, τι άποψη έχετε, τι άποψη έχει η Προεδρία για την ε, σήμανση και όχι μόνο του κλόνου του ιδίου αλλά και των απογόνων του. Γιατί η Κομισιόν θεωρεί πως πρέπει να σημαίνεται μόνο το όντω κλωνοποιημένο ζώο και όχι η απογονή του, κάτι το οποίο έχει ζητήσει και το, κάτι το οποίο έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο. Βεβαίως Κατάγεστε από μια χώρα που στο πλαίσιο της κρίσης αντιμετωπίζει δυσκολίες και η γεωργία, ειδικά όσον αφορά τις μικρές εκμεταλλεύσεις, ε, από τις οποίες υπάρχουν πολλές στην ε, χώρα σας. Θα θέσετε ξανά το θέμα του πώς θα ληφθούν υπόψη ειδικά αυτές οι μικρές εκμεταλλεύσεις στη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο ε, δηλαδή πρέπει και οι άνθρωποι αυτοί να ε, μπορούν ε, να βγάζουν το, το βιός τους, να συνεχίσουν να, υπάρχουν και ας είναι και μικροί αγρότες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φετσκόψκι τώρα και κατόπιν ο κύριος Νίκολς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ που παρουσιάσατε τους στόχους της ελληνικής προεδρίας. Πράγματι, πρόκειται για μια ακόμα τυπική προεδρία. Θα ολοκληρώσουμε και ένα μεγάλο κύκλο του κοινού μας έργου σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής και τον προϋπολογισμό. Όμως, πολλές αποφάσεις έχουν ήδη ληφθεί και θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αυτή η Προεδρία δεν ε, αντιμετωπίζει και πάρα πολλές δυσκολίες γιατί τα μεγαλύτερα καθήκοντα έχουν ήδη ολοκληρωθεί και τα καινούργια δεν έχουν εμφανιστεί ακόμη στο προσκήνιο. Όμως, ίσως αυτή να είναι η κατάλληλη στιγμή να προβληματιστούμε γιατί η ελληνική προεδρία έχει την ευκαιρία να ξεκινήσει τη συζήτηση σε μια σειρά θεμάτων που θα καταστούν σημαντικό για το επόμενο κοινοβουλευτική θητεία. Και κάποιοι από εμά θα ασχολούνται με τα θέματα αυτά στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο και σίγουρα θα πρέπει να συνεχιστεί συζήτηση για τα θέματα αυτά. Υπάρχουν αρκετά θέματα που ζητούν την προσοχή μας. Παραδείγματο χάρη, ένα θέμα που δεν κατορθώσαμε να λύσουμε πλήρως ή μπορώ να πω ότι αποτύχαμε μάλλον να επιλύσουμε το ζήτημα αυτό κατά τη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου. Και εννοώ τις πολύ μεγάλες διαφορές ε, μεταξύ των άμεσων πληρωμών στα μεμονωμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από ό,τι καταλαβαίνω, εσείς εκπροσωπείτε ένα κράτος μέλος που δεν μπορεί να παραπονεθεί γι' αυτό όμως ε, πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και αφορά κυρίως τα νέα κρατημέλη. Εμείς ε, αισθανόμαστε ως αντικείμενο διάκρισης ε, σε ό,τι αφορά τις άμεσες ενισχύσεις. Και το λέω αυτό ως μέλος πολιτικής ομάδας που πρότεινε οι άμεσες ενισχύσεις, τις άμεσες ενισχύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα έχουμε πληρωμές που δεν βασίζονται τόσο στην παραγωγή όσο στην έκταση. Και εμείς ε, θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν τόσο μεγάλες αποκλήσεις ε, σε ό,τι αφορά αυτές τις πληρωμές. Πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση, αλλά έχουμε και άλλα θέματα ε, σημαντικά, όπως είναι οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί ή η ευημερία των ζώων υπάρχει ένα θέμα έλλειψης διαφάνειας σε κάποια θέματα όπως η κλωνοποίηση. Το αναφέραν και οι συνάδελφοι. Έτσι λοιπόν αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα προς συζήτηση για αυτή την Προεδρία. Πρόκειται για μια Προεδρία η οποία θα μας καθοδηγήσει προς τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο. Ίσως λοιπόν αυτή η Προεδρία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, σε αυτό το πνεύμα δεν χρειάζεται να ε, μπει μια τελεία κατά κάποιο τρόπο γιατί τίποτα δεν θα συμβαίνει στο Κοινοβούλιο. Δηλαδή από τα μέσα Απριλίου και μετά δεν θα έχετε συνομιλητές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όμως εγώ νομίζω ότι μπορούμε να σκεφτούμε τώρα εδώ ποιες είναι οι για το μέλλον. Ευχαριστώ. Bardzo dziękuję. W tej chwili proszę o zabranie. Ευχαριστώ. Η κυρία Πατράου παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω ευχαριστώντας τον κύριο Υπουργό για την παρουσία του εδώ και θα ήθελα να εκφράσω και την υποστήριξή μου όχι μόνο στο πρόγραμμα που μας παρουσίασε, για την ελληνική προεδρία στον τομέα της γεωργίας, αλλά εγώ άκουσα με πολύ μεγάλη ικανοποίηση πολλά από όσα μας ανέφερε εδώ και φυσικά θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία και στο κοινό μας σχεδίο Ευρωπαϊκής Οικοδόμησης. Αναφερθήκατε σε κάποια θέματα που είναι πολύ σημαντικά για μένα. Το πρώτο είναι ακριβώς ο γαλακτοκομικός τομέας. Είπατε ότι είναι απαραίτητο να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα της εφαρμογής ε, του πακέτου στο γαλακτοκομικό τομέα. Εγώ μπορώ να πω ότι έχουμε πάρα πολύ λίγα στοιχεία προς αξιολόγηση αυτή τη στιγμή, γιατί σε πολλές χώρες μόλις άρχισε να εφαρμόζεται. Επίσης, αναφερθήκατε στο αν θα αρκέσουν τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα για τη διαχείριση των κρίσεων. Εμείς γνωρίζουμε ότι στο γαλακτοκομικό τομέα είναι κυκλικές οι κρίσεις και επομένως ε, έχουμε ε, μια θετικής ε, περίοδου πάντοτε να ακολουθεί μια αρνητική στο γαλακτοκομικό τομέα και εγώ τολμώ να πω εδώ ότι εμείς δεν είχαμε de facto μία μεταρρύθμιση του γαλακτοκομικού τομέα στην ε, ΚΟΑ. Δηλαδή είχαμε το πακέτο για το γαλακτοκομικό τομέα και τον περασμένο Σεπτέμβριο η Κομισιόν επρόκειτο να παρουσιάσει νέα μέτρα για να ρυθμίσει το γαλακτοκομικό τομέα. Η αλήθεια είναι ότι το μόνο που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι η βεβαιότητα του τέλους των ποσοστώσεων για το 2015 και μία δέσμη μέτρων που ε, είναι ανεπαρκής και πολλές φορές που δεν αρμόζουν στους, στον τομέα, κυρίως στις χώρες του Νότου. Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε αρκετό γάλα στην Ευρώπη, δεν θα λείψει. Όμως ε, ε, αυτές οι περιοχές ε, που παράγουν συνήθως, όπως συμβαίνει στη χώρα μου, είτε στις Αζόρες που είναι άκρως απομακρυσμένη περιοχή, είτε στη Βόρεια Πορτογαλία, είναι οι περιοχές αυτές σε πολύ μεγάλο κίνδυνο με το τέλος των ποσοστώσεων. Έτσι λοιπόν, επειδή μιλήσατε για το γαλακτικό τομέα και για τις μειονεκτικές περιοχές, θέλω να ρωτήσω τι θα κάνει η Προεδρία σας σε σχέση με αυτό το τομέα ο οποίος απασχολεί τόσους γεωργούς και κτηνοτρόφους στην Ευρώπη και βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο αηφορίας, βιωσιμότητας. Και Έχουμε και το θέμα της άνησης ε, κατανομής ε, ε, των μεταρρυθμίσεων στην αγροδιοτροφική αλυσίδα. Εμείς ε, ξέρουμε ότι ακόμη και αν είχαμε κάποια ε, μέτρα όταν εμείς δεν εγγυηθούμε τη δίκαιη κατανομή σε όλο το μήκος της αλυσίδας δεν θα έχουμε μία γεωργία στην Ευρώπη ισορροπημένη. Και από την άλλη όψη του νομίσματος ε, ε, θα πρέπει να έχουμε μία ίση νομή στην διατροφική αλυσίδα. Δυστυχώ, σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα μέτρα ήταν πολύ ε, αδύναμα και δεν είχαν επιπτώσεις σημαντικές και γι' αυτό εγώ φοβάμαι αν δεν κάνουμε σημαντικά βήματα σε αυτό το τομέα η ίδια μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής δεν θα έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Κύριε Υπουργέ, είχατε και την ευαισθησία να αναφερθείτε στις μικρές, στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Τώρα, στο 2014, έχουμε το Διεθνές Έτο της Οικογενειακής Γεωργίας και είναι πολύ σημαντικό να δούμε αυτό τον ιστό γεωργών που είναι κύρια υπεύθυνοι και έχουν μια στενή σύνδεση με τη γη, ε, μια σχέση στοργής ε, πολιτισμού, ιστορίας ε, με τη γη. Πρόκειται πραγματικά για την οικογενειακή γεωργία η οποία διασφαλίζει τη συνοχή στην οποία αναφερθήκατε και διασφαλίζει και τις θέσεις εργασίας. Υπάρχουν πρωτοβουλίες από την πλευρά της Προεδρίας σας σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη αυτού του σχεδίου που είναι ένα παγκόσμιο σχέδιο και είναι ένα ευρωπαϊκό σχέδιο σε ό,τι αφορά τον κλάδο της οικογενειακής γεωργίας. Θα ήθελα να τοποθετηθείτε και σε αυτό. Και μια τελευταία ερώτηση θέλω να θέσω. Αναφερθήκατε στα νησιά. Εγώ θα αναφερόμουν στο ΠΟΖΕΙ, που είναι ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα γεωργίας για τις ε, άκρες απομακρυσμένες περιοχές ε, και θα βρεθεί στο τραπέζι του Συμβουλίου και της Κομισιόν τους επόμενους μήνες ε, και θα έχουμε σύντομα ένα νέο κανονισμό ΠΟΖΕΙ. Το ΠΟΖΕΙ είναι ένα πρόγραμμα που έχει λειτουργήσει πολύ καλά και το μόνο πρόβλημα που έχει είναι ότι δεν ήταν επαρκής η χρηματοδότηση, γιατί ε, πάντοτε είναι λυπής η χρηματοδότηση. Εξαντλήθηκε όμως όλες οι μελέτες δείχνουν ότι στις άκρες μικρές περιοχές έχει λειτουργήσει πολύ καλά το πρόγραμμα. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, και είναι τελευταία ερώτηση, Ποια είναι η θέση της ελληνικής προεδρίας σε σχέση με τα προγράμματα ΠΟΖΕΗ που αυτή τη στιγμή ε, είναι ανοιχτά και φοβούνται οι άνθρωποι ε, σε αυτές τις περιοχές ότι οι μεταρρυθμίσεις που θα γίνουν θα είναι ζημιογόνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στην Ελληνική Προεδρία, κυρίως στον τομέα της Γεωργίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Ράνς Γκαρσία. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Υπουργό που και καθήκοντα Πρόεδρο και που μας εξήγησε εδώ τις προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας. Έχουμε τώρα τον κανονισμό που συζητείτε εδώ. Εσείς είπατε ότι αποτελεί προτεραιότητα για την ελληνική προεδρία. Επίσης, ανακοινώσατε ότι θέλετε να πετύχετε μια συμφωνία κατά τη διάρκεια της αιτίας σα. Εμεί, ε, ω Κοινοβούλιο θα ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας τον Απρίλιο και έχουμε τις εκλογές τον Μάιο και επομένω μας πιέζει ο χρόνος. Εσείς πιστεύετε ότι είναι δυνατόν να πετύχετε μια συμφωνία με το Κοινοβούλιο από τη στιγμή που θα ψηφιστεί το Μάρτιο στην Επιτροπή Άγκρη και τη Ολομέλεια του Απριλίου. Γιατί θα έπρεπε να ζητήσονται όλοι στην Επιτροπή για να το διαπραγματευτώ μαζί σας πριν από την ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Jako ostatni zabierze głos pan poseł. Ωραία. Ο κύριος Γιάρ. Ε, ναι, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Έχω μία σύντομη ερώτηση Είπατε σωστά πως το κέντρο της ε, δουλειάς σας θα βρίσκεται η σωστή εφαρμογή της μεταρρύθμισης κοινής γεωργικής πολιτικής, ε, ε, πράξη κατεξιοδότηση και τα λοιπά. Αλλά στο θέμα της μείωσης της γραφειοκρατίας, δεν ξέρω τι έχουμε κάνει, γιατί η μείωση της γραφειοκρατίας για τους αγρότες δεν έχει προχωρήσει. Διαπιστώνουμε πως με κάθε μεταρρύθμιση ε, το σύστημα γίνεται πιο γραφειοκρατικό για τον αγρότη. Και πρέπει να ομολογήσω και να κάνω την αυτοκριτική μας πως και εμείς οι ευρωβουλευτές ε, φταίμε. Τα κάνουμε τα πράγματα όλο και πιο πολύπλοκα. Οπότε θα ε, σας έλεγα να προσπαθήσετε πως τουλάχιστον για τους αγρότες η μεταρρύθμιση να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο γραφειοκρατική. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, Υπουργέ. Θα σας δώσω τώρα το λόγο για να κάνετε κάποιες ε, σύντομες ε, παρατηρήσεις. Θα ήθελα πέρα από αυτά τα ερωτήματα να σχολιάσετε και τις επιπτώσεις της κρίσης επί του γεωργικού τομέα, αν έχετε την καλοσύνη. Νομίζω δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις από τους συναδέλφους. Ε, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ και πάλι κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις όλες τις επιμέρους ερωτήσεις που τέθηκαν και θα αρχίσω από την πρώτη που τέθηκε από αρκετούς ε, βουλευτές και αφορούσε τα θέματα των κατεξουσιοδότηση πράξεων και τι θα κάνουμε ε, στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Όπως έχω πει, η έγκριση των κατεξουσιοδότηση πράξεων είναι κοινή επιδίωξη τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου και θεωρώ είναι και του Ευρωκοινοβουλίου προτεραιότητα, ώστε να μην προκύψουν εμπόδια για την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ από την 1η Πρώτου του 2015. Αυτό είναι ζητούμενο και από τα τρία μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Προεδρία για να βοηθήσει προς το σκοπό αυτό οργάνωσε ήδη στις 13 Ιανουαρίου συζήτηση στο ειδικό στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας για το θέμα αυτό και οι αντιπροσωπείες των κρατών μελών εξακολουθούν να έχουν ανησυχίες. Αναμένουμε τα αποτελέσματα της ενδοϊπηρησιακής διαβούλευσης της Επιτροπής και τα νέα κείμενα των κατεξουσιοδότηση πράξεων που θα υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Συμβούλιο και στο Ευρωκοινοβούλιο. Ευελπιστούμε, όπως τόνισα και στην ομιλία μου, ότι θα έχουν ληφθεί υπόψη τόσο οι απόψεις των κρατών μελών, δηλαδή το, του Συμβουλίου, όσο και οι ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι δεν θα υπάρξουν κίνδυνοι απόρριψη των νέων αυτών κειμένων. Οι Ευρωπαίοι γεωργοί χρειάζονται ένα σταθερό περιβάλλον, αυτό τονίστηκε από όλους σχεδόν, προκειμένου να προγραμματίσουν την παραγωγή και τις επενδύσεις τους. Τα κράτη-μέλη χρειάζονται επίσης τους οριστικούς και πλήρεις κανόνες για να προχωρήσουν στις κρίσιμες για τη βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα επιλογές τους, όπως ο σχεδιασμός των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης, οι μεταφορές πόρων μεταξύ των δύο πυλώνων, οι συνδεδεμένες ενισχύσεις κλπ. Γνωρίζετε ότι σε περίπτωση τυχόν απόρριψης τώρα δεν υπάρχει δυνατότητα επανεποβολής των προτάσεων πριν την ανάληψη των καθηκόντων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό τη νέα τη σύνθεση. Πιστεύω ότι Όλοι θα ακούσουν τα συγκεκριμένα μηνύματα και όλοι θα αναλάβουν τις ευθύνες τους γι' αυτό. Ως προς το κομμάτι των, ε, της ασφάλειας των ζώων, των φυτών και των, την ασφάλεια του αγροδιοτροφικού τομέα. Τονίστηκε ιδιαίτερα το κομμάτι του φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού. Η ελληνική Προεδρία, σας είπα, θα εργαστεί από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα ανοίξει το δρόμο για την επίτευξη μιας μελλοντικής συμφωνίας. Γνωρίζουμε πολύ καλά τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από ορισμένους βουλευτές, αλλά και των πολιτικών ομάδων σχετικά με τις διάφορες προκλήσεις που προτείνονται στην πρόταση. Το Συμβούλιο εξετάζει προσεκτικά την πρόταση αναφορικά και με τις επιπτώσεις και τις συνέπειές της. Οι εκτιμήσεις αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για μια τέτοια πρόταση η οποία έχει ως στόχο να εξυγχρονίσει και να απλουστεύσει ένα μεγάλο αριθμό λεπτομερών τεχνικών μέτρων που ισχύουν εδώ και πολλά χρόνια. Βέβαια αρκετή, απαιτείται, συμφωνώ, αρκετή δουλειά ακόμη ώστε να πετύχουμε σαφείς κανόνες και νομική ασφάλεια συμπαραλαμβανομένων και εκείνων που θα καθορίσουν στη συνέχεια που θα καθοριστούν στη συνέχεια με τις εξουσιοδητικές και εκτελεστικές πράξεις. Τώρα, ένα επίσης θέμα που τέθηκε και αφορά το θέμα των, ε, των κλώνων και της κλωνοποίησης των ζώων. Όπως είπα, είναι ένα σημαντικό θέμα. Η συζήτηση για τις προτάσεις αυτές δεν έχει ξεκινήσει ακόμα στο πλαίσιο του Συμβουλίου και των προπαρασκευαστικών οργάνων του. Δεν υπάρχουν πολλά που μπορούμε να πούμε σε αυτό το στάδιο για το περιεχόμενο. Η Προεδρία σκοπεύει να ξεκινήσει όμως τη συζήτησή του στα όργανα του Συμβουλίου. Σε ό,τι αφορά το θέμα των ε, τα βιολογικά. Το βιολογικό σύστημα παραγωγής είναι ένα σημαντικό παραγωγικό σύστημα καλλιέργειας, ενδιαφέρει πάρα πολλούς τους καταναλωτές που θέλουν να έχουν ένα τέτοιο παραγωγικό σύστημα και προτιμούν τα προϊόντα του. Πολλά κράτη-μέλη είναι υπέρ της απλοποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας. Η Επιτροπή επίσης αναγνωρίζει ότι η υφιστάμενη νομοθεσία περιέχει μειονεκτήματα που πρέπει να επαναξεταστούν η ελληνική προεδρία καλωσορίζει αυτή την πρόταση της Επιτροπής να παρουσιάσει την νομοθετική της πρόταση το Μάρτιο, όπως εκτιμάται τουλάχιστον, και είναι έτοιμη να ασχοληθεί με την νέα αυτή πρόταση και να την προχωρήσει όσο μπορέσει. Ό,τι βήματα κάνουμε θα είναι προς, το, προς όφελος και της βιολογικής γεωργίας και των Ευρωπαίων καταναλωτών. Σε ό,τι αφορά το θέμα του γαλακτοκομικού τομέα που τόνισα και ε, αναφέρθηκε επίσης. Ανέφερα ήδη ότι θα εξετάσουμε όλα τα αποτελέσματα της εφαρμογής του γαλακτοκομικού πακέτου που θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο του 2004. Ενώ έχουμε ήδη προγραμματίσει συζήτηση για το πρώτο τρίμηνο του 2014 σχετικά με το μέλλον του τομέα αυτού. Σας θυμίζω ότι πολλά από τα θέματα θύχθηκαν στο συνέδριο που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2013 και αφορούσαν μέτρα για την αντιμετώπιση των, και τα, προβλήματα, τα απορίσματα αυτού του συνεδρίου παρουσιάστηκαν στο Συμβούλιο μας τον περασμένο Δεκέμβριο. Μια και αφορούσαν όπως είπα τα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων σχετικά με τη διατήρηση της παραγωγής, ιδιαίτερα στις μειονεκτικές περιοχές που κι εσείς αναφέρατε. Καθώς και στην αξιοποίηση των εργαλείων της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής, ειδικά για τις περιοχές αυτές ένας από τους σημαντικότερους στόχους της νέας κοινή αγροτικής πολιτικής είναι η διατήρηση της παραγωγικής γεωργίας σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές όπως και στις εξόχως απόκεντρες που αναφερθήκατε. Είναι νομίζω περιττό να επαναλάβω και να τονίσω ότι το γάλα είναι ένα σημαντικό τομέα. Θα κάνουμε συζήτηση προς ανατολισμού στο μέσο της Προεδρίας μας Αναμένουμε και την έκθεση της Επιτροπής όπως τόνισα τον Ιούνιο. Είναι τόσο μεγάλο το θέμα που ε, η εξέτασή του θα απασχολήσει και το επόμενο κοινοβούλιο, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Σε ό,τι αφορά τα θέματα της βιοτεχνολογίας και ιδιαίτερα το θέμα του καλαμποκιού στο οποίο αναφερθήκατε. Το καλαμπόκι με αριθμό 1507. Γνωρίζετε καλά ότι από το 2010 η Ευρώπη δεν έχει γκρίνει καμιά γενετική τροποποίηση σε φυτικές ποικιλίε φυτών για καλλιέργεια. Η τελευταία ήταν η πατάτα αμφλόρα, σας θυμίζω ότι της οποίας η έγκριση ακυρώθηκε από το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 13 Δεκεμβρίου του 2013, άρα δεν υπάρχει πλέον η μόνη εγκεκριμένη καλλιέργεια παραμένει το καλαμπόκι της Μονσάντο, Μονσάντο 810, της οποίας μάλιστα εκρεμεί η ανανέωση της έγκρισης εδώ και αρκετά χρόνια. Τώρα, σε ό,τι αφορά το καλαμπόκι της παίονιρ 1507. Αφότου το σχέδιο απόφασης κατατέθηκε στην Επιτροπή μετά την γνωστή δικαστική απόφαση και απασχολεί πλέον την Προεδρία, ακολουθήσαμε τη γνωστή διαδικασία με την εξέταση στο Κορεπέρ. Σήμερα εξετάζεται σε τεχνικό επίπεδο και την Παρασκευή πάλι στο επίπεδο Κορεπέρ θα δηλωθεί η πρόθεση ψήφου των κρατών μελών. Να δούμε δηλαδή αν τα κράτη-μέλη τοποθετούνται με τον ίδιο τρόπο όπως τοποθετήθηκαν και στο παρελθόν ή έχει αλλάξει κάτι. Η διαδικασία είναι πολύ συγκεκριμένη επιβάλλεται όπως ξέρετε καθορίζεται ήδη από τα, τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του Συμβουλίου και η Προεδρία δεν έχει καμιά δυνατότητα να παρεκκλίνει από αυτούς τους κανόνες. Δεν ξέρω αν άφησα κάποιο από τα θέματα αναπάντητα, αναφέρθηκα. Να γνωρίσω κάτι που είναι το για την πρωτοβουλία Ποσέη για τα νησιά, επαναλαμβάνω και πάλι, γνωρίζετε πάντως, μιλώντας τώρα ως υπουργό της Ελλάδος, ότι έχουμε κοινέ ευαισθησίες για τις, αξέχουσες, για τις εξαιρετικά αυτές μικρές και απόμακρες περιοχές. Τέλος, ήθελα να πω κάτι και να κλείσω με αυτό κύριε Πρόεδρε, γιατί τονίστηκε ήδη, μια και αναφέρομαι μάλιστα και στη χώρα μου, να πω ότι η χώρα μου παρά το ότι είναι μια μικρή έκταση χώρα, εν τούτης, έχει μια ποικιλομορφία των παραγωγικών της συστημάτων, δεν είναι ίδια η γεωργία ενός μικρού νησιού από ότι είναι η γεωργία στα βουνά της Ελλάδος και αυτή η ποικιλομορφία των αγροπεριβαντολογικών συστημάτων της αντικατοπτρίζεται και στον πλούτο και την ποικιλομορφία και την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων. Πιστεύω ότι αυτό που χαρακτηρίζει τη χώρα μου χαρακτηρίζει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει ποικιλομορφία αγροτικών συστημάτων, ποικιλομορφία εξαιρετικών προϊόντων. Επειδή πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα στρατηγικό πλεονέκτημα της Ευρώπης, στο άτυπο συμβούλιο που θα γίνει στη χώρα μας στα πλαίσια της ελληνικής προεδρίας μεταξύ 4ης και 6 Μαΐου το θέμα της συζήτησης στο Συμβούλιο μας θα είναι αυτό. Πώς αυτή, αυτό, αυτή η ποικιλομορφία των παραγωγικών συστημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μετατραπεί σε ένα από τα σημαντικά της στρατηγικά πλεονεκτήματα. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε, Υπουργέ, για τις πληροφορίες που μας παρουσιάσατε. Σας ευχαριστούμε για όλες τις απαντήσεις που δώσατε. Θα σας ευχηθούμε καλή επιτυχία για την Προεδρία, καλή δουλειά. Όντως, δεν είναι χαρακτηριστική η Προεδρία λόγω των ιδιαιτεροτήτων της, ε, της χρονικής στιγμής, όπως προαναφέραμε. Πρόκειται για μια περίοδο επίσης περισυλλογής για τη μελλοντική πορεία. Δεν θα θέλαμε λοιπόν να είναι μια μεταβατική περίοδος. Θέλουμε να ληφθούν δράσεις που θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη μελλοντική πορεία της Γεωργίας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για όλες τις αναφορές που κάνατε για την κατάσταση της γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ότι η κοινή γεωργική πολιτική πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις γεωγραφικές, ε, κλιματικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες ε, της Ευρώπης. Εξυπακούεται ότι το έργο είναι πάρα πολύ δύσκολο να ορίσουμε μια κοινή πολιτική. Δίχως όμως κοινή πολιτική δεν έχουμε εγγυημένο μέλλον. Θα πρέπει λοιπόν να συνυπολογιστούν οι διαφορές μας που αφενός είναι κάτι θετικό αφετέρου δημιουργούν και προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση θα θέλαμε και πάλι να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία στην Επιτροπή μας. Καλή δουλειά και ολοκληρώνουμε το πρώτο τμήμα της σημερινής μας ε, συνεδρίασης. Ε, θα διακόψουμε για ένα λεπτό για να αποχαιρετήσουμε τον Υπουργό. Thank you, for your Υπότιτλοι AUTHORWAVE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 No, no. I know. That's from the third expert. Yes, I know, I know. Thank you. Prosimy o zajmowanie miejsc. Proszę Państwa, przechodzimy do... Αγαπητοί συνάδελφοι, να περάσουμε τώρα στο τελευταίο σημείο της ημερησίας διάταξης. Έχουμε ένα εργαστήριο, ένα σεμινάριο με θέμα μέτρα σε επίπεδο καλλιεργειών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη Γεωργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σεμινάριο προετοιμάστηκε από το υπόλοιπο Β, από το τμήμα πολιτικής και οργανώθηκε κατόπιν αιτήματος της δικής μας Επιτροπής και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονες για το έργο τους. Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι κλιματικές αλλαγές είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο συνεχώς ε, απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες προκλήσεις ε, και στον κλάδο της γεωργίας ε, και πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή τα επόμενα έτη. Υπάρχουν πολύ μεγάλες προσδοκίες και για το σημερινό σεμινάριο έχουμε εμπειρογνώμονες στο ζήτημα αυτό. Θα ήθελα να καλωσορίσω τους τρεις προσκεκλημένους μας, τον κύριο Χόρντι Ντομίνγκο, τον κύριο Νικόλα Μεταγέ και τον κύριο Σιλβάν Πελερά. Θα ακούσουμε τους εμπειρογνώμονες. Δεν ξέρω με ποια σειρά σκοπεύετε να πάρετε το λόγο. Ίσως θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε τη σειρά που έχω εδώ και καταρχήν Θα μπορούσαμε να ακούσουμε τον κύριο Ντομίνκο. Και νομίζω ότι πρέπει να έχετε κατά νου σας τη διάταξη αυτή. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Eh, Ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόσκληση να παρουσιάσει τα αποτελέσματα των εργασιών μας. Ο στόχος ε, της μελέτης που παρουσιάζεται εδώ και που έχετε στα χέρια σας είναι να δώσουμε μια αντικειμενική και πλήρη ανάλυση για τις ε, επιλογές μείωσης των σε επίπεδο εκμετάλλευσης. Επίσης, θέλουμε να διευκολύνουμε τη λήψη αποφάσεων από την πλευρά των ευρωπαϊκών και εθνικών αρχών σε σχέση με τη νέα μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και την καταπολέμηση της κλιματική αλλαγή. Επομένως, συνειδητοποιούμε ότι οι ακόλουθες μεταρρυθμίσεις της ΚΑΠ ήθελαν να αντιμετωπίσουν σημαντικές προκλήσεις σε επίπεδο περιβάλλοντος και εδώ η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ υποθέτει μία μεγάλη ευκαιρία για το μετριασμό των κλιματικών λαγών. Όπως θα εξηγήσουμε τα επόμενα λεπτά και υπάρχει δυνατότητα συμπερίληψης μέτρων με σημαντική δυναμική, σημαντική δυνατότητα μετριασμού και στον πυλώνα 1 και στον πυλώνα 2. Ο τελικός αντίκτυπος των μέτρων αυτών είναι αβέβαιος ακόμη και εξαρτάται από το αν τα μέτρα προτείνονται στην έκθεση αυτή τελικά θα αναπτυχθούν ε, στα πλαίσια των προποθέσεων που έχουν περιγραφεί και αν τα κράτη-μέλη κάνουν προσπάθεια για να τα συμπεριλάβουν ιδίως στο δεύτερο πυλώνα. Αυτή η ευελιξία που έχει δοθεί στα κράτη-μέλη θα είναι ε, κάτι βασικό για να δούμε αν τελικά θα έχουμε πλεονέκτημα ή μειονέκτημα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Αυτή η έκθεση βασίζεται κυρίως στα αποτελέσματα ενός προγράμματος live και βλέπετε εδώ τη δομή του. Έχουμε πέντε εταίρους από τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν εργαστεί για να ε, μπορέσουν να βρουν τα πιο αποτελεσματικά μέτρα σε επίπεδο εκμετάλλευσης. Και εδώ έχουμε αναλύσει τα διάφορα μέσα αξιολόγησης που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, αξιολογήθηκαν με ένα πρακτικό και εφαρμοσμένο τρόπο. Έχουμε πραγματικά δεδομένα από πάνω από 120 ευρωπαϊκές εκμεταλλεύσεις και εδώ συμπεριλαμβάνεται μια μεγάλη γκάμα παραγωγικών συστημάτων. Εδώ, στο στην διαφάνεια αυτή βλέπετε την αξιολόγηση ε, των εκπομπών ε, του που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και ακολουθούμε διεθνή μεθοδολογία. Εδώ μπορείτε να δείτε τις χώρες που εμπλέκονται. Πρόκειται για, τέσσερις, για τις τέσσερις πλέον σημαντικές οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ δέχεται την ποικιλομορφία των παραγωγικών συστημάτων επί των οποίων εργαστήκαμε. Και όπως σας είπα έχουμε χαρακτήρα εφαρμογής. Για κάποια χρόνια συνομιλήσαμε με αυτούς τους γεωργούς και συνεργαστήκαμε μαζί τους και είδαμε ποια είναι η πρόοδος αυτών των εκμεταλλεύσεων σε ό,τι τη μείωση των εκπομπών ανά περίοδο έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα μέτρα αυτά και αφού τέθηκαν σε εφαρμογή αξιολογήσαμε τα αποτελέσματα, την επιτυχία τους δηλαδή και τελικά μεταξύ όλων αυτών των μέτρων καταλήξαμε σε 12 μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν σε αυτούς τους άξονες που βλέπετε. Πρόκειται για μέτρα γεωπονικού τομέα, μέτρα μετριασμού για την κτηνοτροφία και μέτρα που αφορούν την ενέργεια. Και τέλος ε, έχουμε και ένα τέταρτο άξονα που μιλά, ε, το προτείνουμε ε, και λέμε ότι έχουμε γεωπεριβαλλοντικά μέτρα χαμηλού άνθρακα, έναν ευέλικτο μηχανισμό δηλαδή έτσι ώστε οι γεωργοί να μπορούν να εκτελέσουν και να εφαρμόσουν τα μέτρα που θα είναι πιο κατάλληλα για τις δυνατότητές τους και ανάλογα με τους περιορισμούς που έχουν και να δουν ποια μέτρα είναι δυνατόν να εφαρμόσουν στη δική τους εκμετάλλευση. Στη μελέτη που έχετε στα χέρια σας, επίσης, έχει γίνει ένα μικρό βήμα σε σχέση με τα αποτελέσματα του προγράμματος και για κάθε ένα από τα μέτρα που είχαμε στο προηγούμενο σχεδιάγραμμα γίνεται μια τεχνική περιγραφή και τίθενται κάποιοι τεχνικοί στόχοι. Έτσι, εδώ βάσει των τεχνικών στόχων εντοπίζουμε τα παραγωγικά συστήματα που εντάσσονται εδώ και τη δυναμική μείωση ε, των εκπομπών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης ήταν πολύ σημαντικό για μας να εντοπίσουμε τις περιβαλλοντικές συνεργίες, ε, συνέργειες που μπορεί να εφαρμοστούν για το μετριασμό και είναι πολλές οι συνέργειες αυτές. Και ένας άλλος στόχος, ένα άλλο από τα αιτήματα του Κοινοβουλίου, ήταν να εξηγήσουμε σε ποια μέσα της νέας ε, μεταρρύθμισης της κοινή ε, γεωργικής πολιτικής θα ήταν δυνατόν να εφαρμοστούν ε, τα μέτρα αυτά. Διαφορετικά να προτείνουμε εναλλακτικά μέτρα. Επίσης αναλύεται η δυσκολία για τους γεωργούς ως προς την εκτέλεση των μέτρων αυτών, καθώς και η δυνατότητα παρακολούθησης από την πλευρά εθνικών ή ευρωπαϊκών αρχών για την υλοποίηση των μέτρων. Επίσης γίνεται μια ανάλυση του κόστους εφαρμογής ε, καθώς και των περιορισμών. Με όλα αυτά τα στοιχεία καταλήγουμε σε μια ιεράρχηση των μέτρων αυτών και αυτή η ιεράρχηση βασίζεται κυρίως σε τρεις σημαντικές αποφάσεις. Η πρώτη είναι ε, το βελινικές που έχουν τα μέτρα αυτά σε επίπεδο εκμετάλλευση, δεύτερον το κόστος και τρίτον οι δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν οι γεωργοί για την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Εδώ βλέπετε ένα πίνακα, είναι πολύ μικρά τα γράμματα, δεν φαντάζομαι να μπορείτε να το διαβάσετε, απλώς σας το παρουσιάζουμε για να δείτε μια σύνοψη με τι ακριβώς εργαστήκαμε μπορείτε να δείτε εδώ, στα πλαίσια αυτών των μέτρων. Όπως βλέπετε, για κάθε μέτρο εντοπίζεται η δυναμική, ο στόχος που θέλουμε να πετύχουμε και έχουμε και τα υπόλοιπα μέτρα. θα αναφέρω κάποια μέτρα στο γεωπονικό τομέα. Αναφερόμαστε εδώ στο ισοζύγιο αζότου σε επίπεδο εκμετάλλευσης, δηλαδή βελτιστοποίηση του ορυκτού αζότου σε επίπεδο εκμετάλλευσης θέτοντας κάποιους στόχους και κυρίως εξηγώντας ότι πρόκειται για ε, κάτι, μια, μια αξιολόγηση που γίνεται μετά τη σοδιά και όχι πριν τη σοδιά, πριν τη συλλογή της σοδιάς. Δεύτερον, έχουμε την εισαγωγή των ε, λογοφόρων λαχανικών. Τρίτον, την γεωργία συντήρησης, διατήρησης και εδώ θεωρούμε ότι δεν βασίζεται αποκλειστικά ε, σε χρήση μηχανημάτων άμεσης σποράς αλλά σε και σε άλλα μέτρα όπως έχουμε την άμεση σπορά ή ε, τη χρησιμοποίηση προστατευτικών καλλιεργειών ε, κτλ. Αυτό το μέτρο βασίζεται αποκλειστικά αν το βασίσουμε αποκλειστικά στη χρήση μηχανημάτων άμεσης ποράς, χάνουμε μια μεγάλη δυναμική μετριασμού. Και τέλος, έχουμε και τις προστατευτικές καλλιέργειες και σε αυτό το πακέτο βάζουμε και τις ενδιάμεσες καλλιέργειες όπως και τις λεγόμενες catch crops. Τώρα, σε ό,τι αφορά τώρα τα ακτινοτροφικά μέτρα, προτείνουμε εδώ την ε, αποθήκευση της ε, κοπριάς ε, και την ε, κατανομή τη, το σκορπίσμα και επίσης έχουμε και το βιοαέριο σε επίπεδο εκμετάλλευση, τονίζοντας τη, τη σημασία που θα είχε αυτό το μέτρο και δίνοντας προτεραιότητα ε, στη χρήση ε, των ζωικών απορριμμάτων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μέτρα στον τομέα της ενέργειας, μιλάμε για αντικατάσταση του καυσίμου από τη βιομάζα, φωτοβολταϊκή ενέργεια, τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων ε, μέσω διάφορων ε, μοντέλων, αλλά λαμβάνουμε κυρίως ε, υπόψη το γαλλικό μοντέλο και ένα μέτρο που αφορά τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και κυρίως στον γαλακτοκομικό τομέα. Επίσης, επικεντρωνόμαστε σε ένα γεωπεριβαλλοντικό μέτρο που το παρουσιάζουμε ως χαμηλού άνθρακα βάσει της πρακτικής εμπειρίας που προήρθε από το πρόγραμμα όπου διαπιστώσαμε ότι οι γεωργοί όταν τους δίνονται συγκεκριμένες δυνατότητες, ένα συγκεκριμένο μενού θα έχουν δυσκολία να το εκτελέσουν γιατί έχουν περιορισμούς τεχνικού, οικονομικού χαρακτήρα ή προσωπικούς περιορισμούς. Και και το καλύτερο είναι μέσα σε ένα πλαίσιο εργασίας να προτείνουμε μια ευρεία δυνατότητα επιλογών έτσι ώστε ένα μέρος αυτών των μέτρων να τεθούν σε εφαρμογή. Και θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο που θα συνεχίσει τις επεξηγήσεις επικεντρωνόμενος στο τελευταίο αυτό μέτρο. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω και εγώ κάποια συγκεκριμένα αποτελέσματα ε, για τις εκμεταλλεύσεις στα πλαίσια αυτού του προγράμματος. Ε, βλέπετε στις διαφάνειες τώρα ε, τα πορτοκάλια και τα μανταρίνια, την παραγωγή τους στην Ισπανία και τις επιπτώσεις των αερίων του θερμοκηπίου. Βλέπετε πόσο διαφορετικά είναι τα αποτελέσματα ως προς τα αέρια θερμοκηπίου ανά εκτάριο. Τα βλέπετε στον κάθετο άξονα και άλλους δείκτες όπως η κλιματική επίπτωση, ε, δηλαδή αν ε, παραχθεί ε, ποσότητα, ποιες είναι οι επιπτώσεις των αερίων του θερμοκηπίου. Βλέπουμε ότι σε διαφορετικές εκμεταλλεύσεις, ανάλογα με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται, έχουμε διακύμαση από 1 έως 5 σε σχέση με τις επιπτώσεις των αερίων θερμοκηπίου ανά εκτάριο. Ε, βλέποντας λοιπόν το την μπλε ζώνη στη διαφάνεια, ε, κατανοούμε ποιες είναι, ποια είναι τα διάφορα προγράμματα που προτάθηκαν και, τα, και το ευρύ φάσμα μέτρων που κάλυπταν ε, αναφέρονται επίσης οικονομικοί και τεχνικοί περιορισμοί. Κάποια μέτρα ε, υλοποιήθηκαν, ε, τα οποία αναπαρίστανται εδώ με το πράσινο βέλος και αντιστοιχούν σε μία ή περισσότερες δράσεις. Βλέπετε ότι μπορούμε να επιτύχουμε μειώσεις αερίων σημαντικής κλίμακας μετά από την εφαρμογή των μέτρων. Donc, les actions οι δράσεις που εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις είναι επικύλε και εξαρτώνται κάθε φορά από τα συστήματα που χρησιμοποιούνται. Παραδείγματος χάρη, στον πρώτο πίνακα για την παραγωγή πορτοκαλιών ε, μιλάμε για μέτρα, για αζωτούχα λιπάσματα, ε, για την ε, άρδευση με νέα εργαλεία, παραδείγματο χάρη για να αυξήσουμε ή να μειώσουμε την ποσότητα νερού ανά εκτάριο. Ανάλογα το, με το σύστημα λοιπόν, γιατί υπήρχαν τρία διαφορετικά συστήματα για τα πορτοκάλια, με την στάγδιν άρδευση, την επιφανειακή άρδευση ή στη συνέχεια τις βιολογικές εκμεταλλεύσεις, η μόχλευση δεν είναι η ίδια ε, των δράσεων ενώ βλέπετε στον πίνακα ποιο είναι το δυναμικό των μειώσεων. Έχουμε την στήλη για την ε, ε, αποθήκευση του άνθρακα και για τις επιπτώσεις των αερίων θερμοκηπίου και διαπιστώνουμε ότι μπορούμε να επιτύχουμε μείωση 10% για τις επιπτώσεις των αερίων θερμοκηπίου και να διπλασιάσουμε τον αποθηκευμένο άνθρακα. Στη Γερμανία έχουμε εκμεταλλεύσει που ειδικεύονται σε παραγωγή μήλων, διαφορετικές εκτάσεις, ε, διαφορετικά προϊόντα και εκεί εφαρμόστηκαν μέτρα που σχετίζονται με την ε, κατανάλωση των καυσίμων ε, και την χρήση της θερμότητας από τα συστήματα ψήξης για την αποθήκευση των μήλων που μας επιτρέπουν σε, να επιτύχουμε σημαντικό μετριασμό της αναπηπτώσεων των αερίων του θερμοκηπίου. Un autre cas d'étude après les cultures permanentes. Euh, για τα μόνιμα βοσκοτόπια τώρα, θα σας δείξω ε, μια διαφάνεια για τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις για να σας μιλήσω ε, για τη μόχλευση των δράσεων. Εδώ μιλάμε για μεγάλες εκμεταλλεύσεις λοιπόν ε, της Γαλλίας. Πρόκειται για κεκλειμένες εκμεταλλεύσεις μεγάλες κλίσεως και άρα υφίστανται σημαντικά φαινόμενα διάβρωσης. Οι καλλιεργητικές μέθοδοι για τις κεκλειμένες αυτές πλαγιές ουσιαστικά για να αντιμετωπίσουν την διάβρωση προσφεύγουν στην αμυψή σπορά και εναλλάσσουν τις χειμερινές και τις θερινές καλλιέργειες ε, προσπαθώντας έτσι να μειώσουν την διάβρωση ε, χρησιμοποιώντας φυτική κάλυψη κάθε φορά που ε, η απώλεια θρεπτικών υλών από το έδαφος είναι ιδιαίτερα σημαντική λόγω της διάβρωσης. Βλέπουμε επίσης τις προγνώσεις που έχουν γίνει με ένα συγκεκριμένο εργαλείο Βλέπετε λοιπόν ε, πάνω αριστερά το ενεργειακό προφίλ της εκμετάλλευσης και βλέπετε τις ενεργειακές προκλήσεις για τη συγκεκριμένη εκμετάλλευση, αζωτού, χαλιπάσματα, έλεγχος της κατανάλωσης καυσίμων και δεξιά βλέπετε τις επιπτώσεις για την ε, των αερίων θερμοκηπίου και τα ποσοστά αποθήκευσης του άνθρακα. Κατόπιν βλέπετε τα συνδυασμένα μέτρα και όλα τα επιμέρους ε, στοιχεία της ε, ε, γεωργίας διατήρησης, φυτική κάλυψη, παραδείγματος χάρη άμεση σπορά, και μεγάλη σπορά που καλύπτει και τα ψυχανθή βλέπετε για κάθε μία από αυτές τις δράσεις ε, ε, τα αποτελέσματα της μείωσης του αντικτύπου των αερίων του θερμοκήπιου. Για αυτές τις εκμεταλλεύσεις ε, υπάρχει κατανάλωση, μείωση της κατανάλωσης κατά 30% σε σχέση με τον υπόλοιπο τομέα και 30% ε, επίσης μείωση της επίπτωσης των αερίων του θερμοκηπίου. Ε, το σύνολο αυτών των δράσεων μας επέτρεψε να διπλασιάσουμε το ε, ποσοστό της οργανικής ύλης μέσα στο έδαφος καθώς και το ποσοστό του αποθηκευμένου άνθρακα. Με διάφορες καλλιτεργητικές μεθόδους, δεν μιλάμε για μόνιμες καλλιέργειες, μεγάλες καλλιέργειες ή ή βοσκοτόπια ε, μπορούμε να ε, ε, επιτύχουμε μετριασμό της τάξης του 10% στο 40% ε, βεβαίως εξαρτάται από το σημείο εκκίνηση που διαφέρει σε πολύ μεγάλο βαθμό ανάλογα με το είδος των εκμεταλλεύσεων των προϊόντων. Σε τέτοιου είδου ε, προσέγγιση ε, είναι απαραίτητο να κάνουμε και ενεργειακή αξιολόγηση για να καταγράφουμε τις επιπτώσεις των αερίων θερμοκήπιου. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα συγκεκριμένο ενεργειακό εργαλείο για να έχουμε το σημείο εκκίνηση και ε, να μπορέσουμε στη συνέχεια να συναποφασίσουμε με τον Γεωργό ε, τα μέτρα για να μειωθεί ο αντίκτυπο των αερίων θερμοκηπίων. Στα πλαίσια του προγράμματο αναπτύξαμε ένα τέτοιο εργαλείο. Ταυτόχρονα στην Ευρώπη υπάρχουν και άλλε πρωτοβουλίε από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ περιβάλλοντο με το GRC, παραδείγματο χάρη το κοινό ερευνητικό κέντρο Carbon Calculator, ε, υπολογιστή σε άνθρακα παραδείγματο χάρη. Το βλέπετε εδώ, μπορείτε να το ε, κατεβάσετε από, την, από τον ιστότοπό μα. Υπάρχουν και άλλε τέτοιε πρωτοβουλίε, υπάρχουν και εθνικέ πρωτοβουλίε επίση για την περίπτωση των αερίων του θερμοκήπιου, πρέπει να δείτε τις διαφορές ε, περιμέτρου, ε, ε, τις δυνατότητες χρησιμοποίησης αυτών των εργαλείων. Το σημαντικό είναι να γίνει εκτίμηση βάσει της συγκεκριμένη εκμετάλλευσης και μακροχρόνιος προγραμματισμός συνεργασία με τον Γιώργο για να μετριαστούν οι επιπτώσεις των αερίων του θερμοκηπίου. Σε αυτό το πίνακα βλέπετε το σύνολο των μέτρων που αναλύσαμε στην έκθεσή μας ε, προσπαθήσαμε να τα κατατάξουμε, να τα ιεραρχήσουμε ανάλογα με το κόστος. Ε, βλέπετε αριστερά στον άξονα πάνω-πάνω ε, έχουμε ουδέτερο ή και αρνητικό κόστος, δηλαδή με την εφαρμογή τους έχουμε οικονομικό όφελος για τους γεωργούς. Κάτω-κάτω τώρα στην αριστερή στήλη έχετε τα μέτρα για τα οποία υπάρχει ένα υψηλότερο κόστος εφαρμογής στον Έχουμε και ένα δεύτερο δίκτυ για τις δυσκολίες στη δεξιά στήλη, για τις δυσκολίες για τους γεωργούς, ε, δηλαδή μέτρα για τα οποία χρειάζεται πιο έντονη, πιο εντατική παρακολούθηση από πλευράς ε, του γεωργού. Βλέπουμε μία πρώτη ομάδα εκμεταλλεύσεων στο πάνω μέρος του πίνακα, για τις οποίες Έχουμε ευκολία εφαρμογή, αν θέλετε, υλοποίηση από πλευρά ε, των γεωργών. Χρειάζεται λιγότερη παρακολούθηση και ένα σχετικά περιορισμένο κόστος ε, διαφοροποιούνται και κάποια μέτρα σε σχέση με το δυναμικό μετριασμό, παραδείγματο χάρη τα ζωτούχα λοιπάσματα και τα μέτρα που προτείναμε για την παρακολούθηση των εκμεταλλεύσεων μέσω αγροπεριβαλλοντικών μέτρων για να έχουμε δράσεις που ε, παράγουν λιγότερο άνθρακα. Ε, δεύτερη ομάδα εκμεταλλεύσεων ε, και ως προς την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ και την αποθήκευση κοπριάς το αρνητικό είναι ότι είναι μεγαλύτερο το κόστος εφαρμογής, ταυτόχρονα βέβαια είναι πιο ε, φιλόδοξα ως προς τις δυνατότητες μετριασμού. Προκύπτουν και άλλα τρία μέτρα, η φυτική κάλυψη, παραδείγματος χάρη, στα πλαίσια ε, της ε, γεωργίας συντήρησης ή αηφορίας όπως το ορίζουμε στην μελέτη μας και αξιοποίησης των περιτομάτων των ζώων ε, και ε, μέτρα βιοαερίου που μας επιτρέπουν να επιτύχουμε μεγαλύτερο ε, μετριασμό, όμως η εφαρμογή τους είναι πιο περίπλοκη και επισύρουν ένα, μάλλον απαιτούν μια πιο εντατική παρακολούθηση. Ποιες είναι, οι είναι συμπεράσματα της έκθεσής μας. Υπάρχουν ε, ε, δυνατότητες μετριασμού 10 έως 40% για τις επιπτώσεις των αερίων θερμοκηπίου σε επίπεδο ε, φάρμας εκμετάλλευσης μπορούμε να έχουμε πολύ σημαντικά ωφέλη λοιπόν με την εφαρμογή των μέτρων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το γεωργικό τομέα μπορούμε επίσης να έχουμε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία κυρίως ως προς την εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών και κλιματικών μέτρων ε, που θα εφαρμόσει ο Γεωργός για να μειώσει τις επιπτώσεις των αερίων του θερμοκηπίου και πιο εντατική χρήση αζωτούχων λιπασμάτων. Τέλος πάντων, δεν κάναμε συστηματική ανάλυση των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων. Μας φαίνεται όμως ότι μπορούν να αναπτυχθούν σημαντικές ε, συνέργειες ε, ανάμεσα στα μέτρα για την ποιότητα του νερού, για την βιοπικιλότητα. Πολύ πιθανή συνδυασμή λοιπόν. Και ε, από όλα όσα προτείνουμε είναι ξεκάθαρο ότι για να ε, εφαρμοστεί αποτελεσματικά η μεταρρυθμισμένη κυρία γεωργική πολιτική θα πρέπει να είναι ακριβέστεροι οι ορισμοί των μέτρων στα μελλοντικά εργαλεία, ούτως ώστε να αποκομίσουμε τα μέγιστα ωφέλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και είμαστε στη διάθεσή σας για τις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Προτείνω τώρα να ακούσουμε την τρίτη παρουσίαση του κυρίου Πελερά και μετά θα μπορέσουμε να κάνουμε και ερωτήσεις. Συμφωνείτε? Δεν βλέπω καμία αντίρρηση. Οπότε θα δούμε τώρα την τρίτη παρουσίαση και μετά θα τη συζητήσουμε όλες. Mm. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, σα ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να κάνω την παρουσίαση αυτή. Λέγομαι Σιλβάν Παλέρα. Είμαι ερευνητή στο Εθνικό Ίδρυμα Γεωπονικών Ερευνών στη Γαλλία, στο Ίντρα, και θα σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα μιας μελέτης ε, στην οποία συμμετείχαν και 20 συνάδελφοι περίπου και ο στόχος ήταν να εντοπίσουμε μέτρα για να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στον γεωργικό τομέα στη Γαλλία. Ένα σημαντικό αριθμητικό στοιχείο που θα σας παρουσιάσω στο τέλος της παρουσίασής μου είναι το εξής αφορά ένα κατάλογο μέτρων που θα μας επιτρέψουν τη μείωση των εκπομπών στον τομέα της γεωργίας. Τα μέτρα αυτά από τη μια χαρακτηρίζονται από την δυνατότητα, από την δυναμική μετριασμού. Βλέπετε εδώ κατά μήκο. σε εκατομμύρια τόνους, δείξω ότι το που δεν μπορούσαν να αποφευθούν και χαρακτηρίζονται επίσης και από το κόστος του σε ευρώ ανά τόνου διοξιδίου του άνθρακα που αποφεύγεται και το βλέπετε αυτό στον κάθε το άξονα. Το κόστος αυτό μπορεί να είναι αρνητικό αν υπάρχει οικονομικό κέρδος για το γεωργό ή θετικό αν υπάρχει διεθνικό κέρδος. Και εδώ, σε αυτό το γράφημα, θα επανέλθουμε και θα το σχολιάσουμε. Αλλά πριν από αυτό θα σας παρουσιάσω τη μέθοδο που χρησιμοποιήσαμε για να καταλήξουμε σε αυτό το γράφημα. Και το σχέδιό μου θα είναι το εξή. Θα υπενθυμίσω κάποια πράγματα για τις εκπομπές, Αριάν θερμοκηπίου στη Γαλλία. Θα μιλήσω για τη μέθοδο που χρησιμοποιήσαμε για να επιλέξουμε τα μέτρα μείωση των εκπομπών αυτών. Κατόπιν θα κάνω μια συγκριτική ανάλυση της δυναμικής μετριασμού και του κόστου. Και επίση, τέλο, θα απαντήσω στο ερώτημα σε ποιο βαθμό η νέα κοινή αγροτική πολιτική θα μπορούσε ή δεν θα μπορούσε να επιτρέψει την εφαρμογή των μέτρων αυτών, την υιοθέτηση των μέτρων αυτών. τα ετήσια εκπομπές ε, φτάνουν τα 528 εκατομμύρια τόνους διοξιδίου του άνθρακα. Η γεωργία αντιπροσωπεύει περίπου το 20% και περίπου 10% για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό σχετίζεται με τη σημασία της γεωργίας στη Γαλλία και σχετίζεται και με τις γαλλικές ιδιαιτερότητες στην παραγωγή ενέργειας το 20% που εκπροσωπεί η γεωργία κατανέμεται σε 50% δηλαδή στο μισό που οφείλεται σε πρωτοξίδιο αζότου που είναι ένα σημαντικό ισχυρό αέριο εκπομπής και σχετίζεται με τη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων. Κατόπιν 40% σχετίζεται με το μεθάνιο CH4 που εκπέμπεται από τα μερικαστικά ή όταν έχουμε και νόσεις. Και μόνο 10% σχετίζεται με την κατανάλωση ενέργειας ε, ορυκτών καυσίμων στο επίπεδο εκμετάλλευση. Ο στόχος της μελέτης ε, που ανατέθηκε στο ΙΝΡΑ από το Γαλλικό Υπουργείο Γεωργίας και Οικολογίας ήταν να επιλέξει 10 μέτρα που επιτρέπουν τη μείωση των γεωργικών εκπομπών αυτά τα μέτρα θα έπρεπε να οδηγήσουν, ε, να αφορούν γεωργικές πρακτικές όπως η χρήση λιπασμάτων, ε, οι ζωοτροφές, ε, μάλλον η διατροφή των ζώων και δεν θα έπρεπε να οδηγήσουν σε βαθιές αλλαγές του γεωργικού συστήματος και του επίπεδου παραγωγής ή της τοποθεσίας. Έτσι, εξετάσαμε μέτρα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν, παραδείγματος χάρη, σε μείωση υπεραγωγή παραγωγής 10% και ένας ε, άλλος στόχος ήταν να αποστικοποιήσουμε τη δυναμική μετριασμού των αυτών και το κόστος τους για την περίοδο 2010-2030. Για να το πράξουμε αυτό, βασιστήκαμε στη διεθνή βιβλιογραφία που μας επέτρεψε να εντοπίσουμε περίπου 100 υποψήφια μέτρα, τα οποία τα εξετάσαμε σύμφωνα με πέντε κριτήρια την επιλεξιμότητα σε σχέση με τα καθήκοντά μας, με αυτό που είχαμε να κάνουμε, την αναμενόμενη μείωση στο γαλλικό γεωργικό πλαίσιο, τη διαθεσιμότητα της απαραίτητης τεχνολογίας για να τεθούν σε εφαρμογή και των επιστημονικών γνώσεων που θα καθορίζουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών και μέτρα που είναι ακόμα υπό έρευνα δεν επιλέχθηκαν θα μπορούσαν να ήταν ενδιαφέροντα για το μέλλον. Τη δυνατότητα εφαρμογής ε, του μέτρου, δηλαδή και την ε, κοινωνική αποδοχή και τέλος τις συνέργειες ε, ή τους ενδεχόμενους ανταγωνισμούς με άλλους γεωπεριβαλλοντικούς στόχους όπως η του ενδεχομενους ανταγωνισμους με αλλους γεωπεριβαλλοντικους στοχους οπως η προστασια της βιοπικιλότητας, την προστασία της ποιότητας των υδάτων. Αυτό μας επέτρεψε να καταλήξουμε σε τέσσερις μεγάλους ε, μοχλούς, σε τέσσερα μεγάλα σύνολα, αν θέλετε, σε δέκα μέτρα και τα οποία υποαποτελούνται από 26 υπομέτρα. Οι υπολογισμοί που κάναμε φαίνονται εδώ στο διάγραμμα για κάθε μέτρο υπολογίσαμε την ε, δυνατότητα μετριασμού, ανά εκτάριο ή αναμονάδα και το πολλαπλασιάσαμε με την πιθανή βάση του μέτρου σε επίπεδο γαλλικής επικράτειας και αυτό μας ε, οδήγησε στην δυνατότητα υπολογισμού του ενδυνάμει μετριασμού σε τόνους διεξιδίου του άνθρακα ανά εκτάριο μέχρι το 2030. Και βλέπετε εδώ τον οριζόντιο άξονα. Και για καθένα από αυτά τα μέτρα υπολογίσαμε και το κόστος ε, σε ό,τι αφορά το διαφυγόν κέρδος για το Γεωργό και αυτό μας ε, επέτρεψε με την διαιρετική μέθοδο, να δούμε ποιο είναι το κόστος του μέτρου για κάθε τόνο διοξιδίου του άνθρακα που αποφεύγεται να παραχθεί. Και εδώ, αυτό το βλέπετε στον κάθε του άξονα. Έρχομαι τώρα στον κατάλογο των μέτρων και των ε, υπομέτρων που εντοπίσαμε. Το πρώτο μεγάλο σύνολο, ο πρώτος μεγάλος άξονας έχει να κάνει με τη διαχείριση του αζότου, 50% των εκπομπών. Και έχουμε λοιπόν το πρώτο σύνολο μέτρων που έχουν ως στόχο να μειώσουν ε, τη χρήση των συνθετικών αζωτούχων λιπασμάτων χάρη σε πέντε τεχνικά υπομέτρα, δεν θα τα αναφέρω λεπτομερώς, σε ένα δεύτερο μέτρο που έχει ως στόχο να αυξήσει τη χρήση των ψυχανθών ε, και στις εκπεριτροπής ε, καλλιέργεια, στην αμεψισφορά, αλλά και στα βοσκοτόπια, γιατί δεν χρειάζεται εκεί η χρήση ζωτούχων. Ένα δεύτερο μεγάλο σύνολο είναι η, δέσμευση, συγγνώμη, η αποθήκευση του άνθρακα στο έδαφος και στη βιομάζα με ένα μέτρο που σκοπεύει το, την ανάπτυξη του μη οργώματος για να αποθηκευτεί ο άνθρακας στο έδαφος. Ένα ακόμα μέτρο που έχει να κάνει με τις, ε, την ανάπτυξη ενδιάμεσων ε, καλλιεργειών ε, και να έχουμε και κάποιες ζώνες απομόνωσης κατόπιν να αναπτύξουμε την γεωδασοκομεία και έχουμε και κάτι ακόμα που αφορά την βέλτιστη διαχείριση των βοσκοτόπων δεν θα αναφερθώ τώρα σε λεπτομέρειες. Τρίτο μεγάλο σύνολο, η τροφή των ζώων με ένα πρώτο μέτρο που έχει να κάνει με τη μείωση ε, της εκπομπής μεθανίου από τα μυρικιστικά, ε, τροποποιώντας ανάλογα την τροφή τους. Και ένα άλλο μέτρο έχει να κάνει με τη μείωση των ε, της περιεκτικότητας σε άζωτο ε, των κενώσεων των ζώων. Ένα τέταρτο μεγάλο σύνολο είναι η διαχείριση ε, του κεφαλαίου με ένα στόχο που έχει ως στόχο με την μεθανοποίηση την παραγωγή βιοαερίου και με τη χρήση των ε, εκρήξεων. Και θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα ε, τα γεωργικά μηχανήματα κτλ. Και τώρα έρχομαι στη σύγκριση αυτών των διάφορων μέτρων και υπομέτρων. Εκ νέου βλέπουμε αυτό το περιβόητο γράφημα όπου έχουμε 26 επιμέρους μέτρα που έχουμε εντοπίσει και το καθένα φέρει και ένα τίτλο. Αυτά τα 26 μέτρα έχουμε οριζόντια το, τη δυναμική, την ετήσια δυναμική μετριασμού των εκπομπών, δηλαδή πόσο επιτρέπουν να μειωθούν οι εκπομπές που προκαλούν εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε μεγατόνους αναέτος και στον κάθε το άξονα έχουμε το κόστος του μέτρου σε ευρώ ανά τόνο διοξιδίου του άνθρακα που αποφεύγεται να παραχθεί. Και τα μέτρα αυτά ταξινομούνται από το λιγότερο δαπανηρό, αριστερά, προς το πιο δαπανηρό, δεξιά. Δηλαδή τα λιγότερο δαπανηρά μέτρα φέρνουν ε, και χρήματα στο Γιώργο, ενώ τα πιο δαπανηρά είναι αυτά που οδηγούν σε σημαντικό διαφυγόν κέρδος για το Γιώργο. Αυτά βρίσκονται προς τα δεξιά. Τώρα, η πρώτη πληροφορία είναι συνολικό δυναμικό μετριασμού που επιτρέπει το σύνολο των μέτρων αυτών, κάνοντας ε, μία πλουστευτική υπόθεση προσθήκης, αν τα προσθέσουμε δηλαδή, φτάνουμε σε πάνω από 30 εκατομμύρια τόνων διεξιδίου του άνθρακα, αντίστοιχο ένα έτος. Όλο αυτό θα μπορούσε να αποφευθεί αν θέσουμε σε εφαρμογή το σύνολο των μέτρων αυτών. Και υπενθυμίζω ότι μιλάμε για πάνω από 5 εκατομμύρια τόνους εκπομπές στη Γαλλική Επικράτεια το χρόνο. Και η δεύτερη πληροφορία που βλέπουμε εδώ είναι ότι αυτό το δυναμικό μπορούμε να δούμε ότι αποτελείται από τρία τρίτα. Το πρώτο, έχουμε τα μέτρα αρνητικού κόστους, δηλαδή που επιφέρουν κέρδος στο γεωργό. Αν το δούμε εκ του σύνεγγυς, σε αυτή την πρώτη ομάδα βλέπουμε μέτρα που σχετίζονται με τεχνικές με τεχνικές προσαρμογές. Θα έχουμε καλύτερη μια καλύτερη προσαρμογή των μεριδών των ζωοτροφών, μέτρα για τη μόνωση των κτηρίων, δηλαδή μέτρα που επιτρέπουν να εξοικονομήσουμε πόρους, έσοδα και αυτό σημαίνει ότι επιτρέπουν τη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και επιτρέπουν και να έχει και κέρδος ο Γιωργός. Είναι μια κατάσταση από που όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Δεύτερο. Τρίτο. Έχουμε τα μέτρα θετικού κόστους αλλά μετριοπαθέως. Κάτω από 25 εκατομμύρια τόνους να φαίνεται εδώ βρέχουμε την μεθανοποίηση, τη δασοκομεία, τα ψυχανθή. Βλέπουμε μέτρα που χρειάζονται κάποιες επενδύσεις στη μεθανοποίηση, παραδείγματος χάρη, ή οδηγούν σε τροποποίηση του συστήματος καλλιέργεια όταν μιλάμε παραδείγματο χάρη την εγκατάλειψη του αργώματο ε, και την καλλιέργεια ε, πρωτεϊνούχων και κάποια μέτρα μπορούν να οδηγήσουν σε μικρή απώλεια εσόδων, αλλά αντισταθμίζονται από μείωση του κόστους. Δηλαδή έχουμε λιγότερη κατανάλωση καυσίμων όταν δεν οργώνουμε ή σχετίζονται με άλλα προϊόντα παίρνουμε το σχάρι ε, τα εξηλία ή την ηλεκτρική ενέργεια στην περίπτωση μεθενοποίησης. Και αυτό εξηγεί το μέτριο, μέτριο κόστος. Πρέπει εδώ να επισημάνουμε ότι η οικονομική ανάλυση των μέτρων αυτών προφανώς εξαρτάται πάρα πολύ από τον τρόπο υπολογισμού και κυρίως από το αν θα ληφθούν υπόψη ή όχι κρατικές επιδοτήσεις. Παραδείγματος χάρη, το να μην λάβουμε υπόψη την ε, επιδότηση που σημαίνει η φορολογική έκπτωση ε, των καυσίμων στο γεωργικό τομέα ενισχύει το ενδιαφέρον του μειοργώματος. Ενώ αν δεν λάβουμε υπόψη την επιδότηση για την εξαγορά της ηλεκτρικής ανάγκης που προκαλείται από τη μεθανοποίηση, τότε αυτό μειώνει το ενδιαφέρον του μέτρου αυτού. Πάμε στην τρίτη ομάδα είναι τα πιο δαπανηρά μέτρα και το κόστος τους ξεπερνά τα 25 ευρώ ανά τόνο δεξιότητα άνθρακα που αποφεύγεται. Πρόκειται για μέτρα που χρειάζονται ε, κάποιες επενδύσεις, παραδείγματο χάρη, να υπάρχουν πυρσί για να καίμε το μεθάνιο ή παραδείγματο χάρη κάποιους αναστολής νητροποίησης ή πρόσθετες ύλε ε, για τη διατροφή των ζώων ή παραδείγματο χάρη κάποιες ε, ενδιάμεσες καλλιέργειες ή θα πρέπει να έχουμε φράκτες που πρέπει να τους συντηρούμε, όλο αυτό σημαίνει κόστος. Και επίσης εδώ θα βρούμε κάποια μέτρα που μπορούν να οδηγήσουν σε απώλεια παραγωγής, όπως ε, παραδείγματος χάρη έχουμε στις απομόνωσης, γιατί έχουμε λιγότερη τελική συμμέκτηση, μειώνεται λοιπόν, ε, μειώνονται τα έσοδα του γεωργού και όλα αυτά δεν επιφέρουν πρόσθετα προϊόντα που θα μπορούσαν να, να τεθούν στην αγορά. Προσοχή λοιπόν, το κόστος των μέτρων αυτών εξετάστηκε σχετίζοντάς το μόνο με τους τόνους διοξίδου του άνθρακα που φεύγονται. Όμως ε, ε, κάποια μέτρα όπως οι φράκτες ή οι ζώνες επομόνωσης ε, δεν έχουν μόνο ενδιαφέρον για τη μείωση των εκπομπών, χρησιμοποιούνται και για άλλους σκοπούς, προστασία της βιοπικιλότητας, βελτίωση της ποιότητας των υδάτων κτλ. Και περνάω τώρα στο τελευταίο μέρος της παρουσίασης. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε αυτά τα ερωτήματα. Ποια είναι τα μέσα της νέας κοινή γεωργικής πολιτικής που θα μπορούσαν να ευνοήσουν την υιοθέτηση των μετρών αυτών. Όπως ξέρετε, πελετραπομένα η νέα ΚΑΠ έχει εισαγάγει τρία μέτρα που αφορούν το πρασίνισμα, την ε, προστασία των μόνιμων ε, βοσκοτόπων, την υποχρέωση της ε, ποικιλότητα σε ό,τι αφορά τι καλλιέργειε και την δημιουργία ζωνών οικολογικού ενδιαφέροντος και ε, μια έννοια πρασινίσματος, green equivalency, έχει εισαχθεί για να ευνοηθούν ορισμένες πρακτικές. Στον πίνακα αυτό έχω βαλθεί στα τρία μέτρα πρασινίσματος της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής με τα 10 μέτρα που εντοπίσαμε στη γαλλική μελέτη για τη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου. Βλέπετε κάποιες συγκλήσεις εδώ. Την προστασία των μόνιμων δοσκοτόπων. Φυσικά αυτό συνδέεται με το μέτρο της βελτιστοποίησης της διαχείρισής τους. Η κυκλομορφία των καλλιεργείων θα μπορούσε να ευνοήσει τα ψυχανθή αλλά θα το ξαναδούμε αυτό το θέμα αργότερα. Και επίσης έχουμε και τη δημιουργία περιοχών οικολογικού ενδιαφέροντος που θα έπρεπε να ευνοήσει τη δημιουργία τέτοιων ζωνών απομόνωση κτλ. Τώρα, αν το δούμε εκ του σύνεγγυς, η επαγόρευση που θα γίνει σε ό,τι αφορά το όργωμα ορισμένων βασκοτόπων αποτελεί προϋπόθεση για τη βέλτιστη διαχείρισή τους, όμως τη μελέτη μας στο μέτρο το σχετικό με τα δοσκοτόπια βασιστήκαμε σε κάποιες συγκεκριμένες τεχνικές, σε κάποια συγκεκριμένη συμπεριφορά, με το χάρη σε ό,τι φορά τη μείωση της χρήσης ζωτούχων λιπασμάτων. Και αυτό δεν θα το ευνοήσει ιδιαίτερα η πράσινη πληρωμή, γιατί ο στόχος είναι να προστατευτούν τα βεσκοτόπια, αλλά όχι να αλλάξει ο τρόπος διαχείρισης. Το μέτρο που αφορά την ε, εναλλαγή καλλιεργειών δεν είναι απαραίτητα δεσμευτικό, έτσι ώστε από μόνο του να ευνοήσει την ανάπτυξη των ψυχανθών. Παρ' όλα αυτά, τα κράτη-μέλη μπορούν να, να χρησιμοποιήσουν μέχρι το 2% του κονδυλίου τους για να υποστηρίξουν αυτές τις καλλιέργειες. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι η κοινή αγροτική πολιτική, αν το επιθυμούν τα κράτη-μέλη, θα ευνοήσει τα ψυχανθή. Και σαφέστατα το μέτρο του πρασινίσματος ε, που αφορά τις ζώνες οικολογικού ενδιαφέροντος θα έπρεπε να ευνοήσει τα μέτρα που εντοπίσαμε στη γαλλική μελέτη δηλαδή τις ζώνες απομόνωσης και τους φράχτες. Και τέλος, αν κατάλαβα όμως καλά, αυτό θα εξαρτηθεί και από την απόφαση των κρατών μελών. Πολλά άλλα μέτρα που εντοπίσαμε στην γαλλική μελέτη θα μπορούσαν να ευνοηθούν μέσω της αρχής ε, του greening equivalency. Δηλαδή, μιλώ για την μείωση της, ε, του εργόματος του ισοδύναμου πρασινίσματος. Και εδώ μιλάμε για την αγροδασοκομεία και για καλλιέργειες αμπελώνων ε, ή οπορώνων. Συνολικά, ίσως και με κάποια αισιοδοξία, η νέα ΚΑΠ θα μπορούσε να ευνοήσει 7 από τα 26 επιμέρους μέτρα που εντοπίσαμε στη Γαλλική μελέτη, αν τα αναφέρω εκ νέου, νέα κοινή αγροτική πολιτική θα μπορούσε να ευνοήσει τη μείωση του οργώματος, της άρρωσης, την γεωδασοκομεία, τις ε, τσαμπελώνε, τις ε, ζώνες των αμπελώνων, τα ψυχανθή, τις ενδιάμεσες καλλιέργειες και τις ε, ζώνες αυτές που αναφέραμε προηγουμένως. Κάναμε έναν υπολογισμό σε επίπεδο γαλλικής επικράτειας, σημείωση που υπολογίστηκε υπό ένα σενάριο που συνδυάζει αυτά τα 7 επιμέρους μέτρα που μπορεί να ευνοηθούν από την ε, νέα ΚΑΠ θα έφταναν σε μείωση 7,5 εκατομμύρια τόνων διοξιδίου του άνθρακα ανά έτος. Και αυτό σημαίνει το 23% της συνολικής μείωσης που υπολογίστηκε για τα 26 μέτρα, για το σύνολο των 26 μέτρα, δηλαδή κάτι λιγότερο από το 1 τέταρτο. Και φαίνεται ότι ο αντίκτυπος της αρχής ε, της πράσινης πληρωμής ε, για το μετριασμό των εκπομπών περιορίζεται από το γεγονός ότι κάποιες γεωργικές πρακτικές, όπως ε, παραδείγματος χάρη χρήση ζωτούχων λοιπασμάτων που προκαλούν πολύ μεγάλες εκπομπές δεν είναι στο στόχαστρο των μέτρων πρεσινίσματος. Και έτσι λοιπόν για να έχουμε πιο φιλόδοξους στόχους θα πρέπει να θέσουμε στο στόχαστρο αυτές τις τεχνικές και μέσω άλλων μοχλών, ίσως μέσω του δεύτερου πυλώνα τα μέτρα πρασινίσματος ευνοούν κυρίως δράσεις που επιτρέπουν την αύξηση της αποθήκευσης ε, του άνθρακα, αλλά δεν έχουν σημαντικά αποτελέσματα επί των ε, ε, εκπομπών διοξιδίου του αζότου στο 50% δηλαδή γεωργικών εκπομπών ή στις εκπομπές του μεθανίου 40% για τι γεωργικέ εκπομπέ, καθώ τα μέτρα του πρώτου πυλώνα δεν έχουν τον αναμενόμενο αντίκτυπο ούτε στη χρήση των πεσμάτων ούτε στην διατροφή των ζώων. Άλλα σχόλια που μπορούμε να κάνουμε και σχεδόν τελείωσα είναι ότι πολλά από τα μέτρα που θα περιμένουμε ότι θα ευνοηθούν από το πρασίνισμα είναι κυρίως μέτρα υψηλού κόστους. Αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι οδηγούν σε μείωση της παραγωγής όπως παίρνουν τους χαριζόνες απομόνωσης ή λόγω του χρόνου εργασίας που χρειάζονται, παίρνουν τους διάμεσες καλλιέργειες ή φράχτες, χρειάζονται χρόνο εργασίας, επομένως υπάρχει κόστος. Να επενθυμίσω, ότι τα μέτρα αυτά, τύπου ζώνες απομόνωσης, φράχτες, διάμεσες καλλιέργειες κτλ, έχουν άλλα, παρουσιάζουν άλλο ενδιαφέρον, προστασία της βιοπικιλότητας, ε, μείωση του κινδύνου της διάβρωσης, ε, προστασία της ποιότητας των δάτων. Δεν μπορούμε λοιπόν να αξιολογήσουμε το κόστος τους μόνο υπό όρους μετριασμού των εκπομπών, γιατί έχουν πολλούς στόχους. Τουλάχιστον αυτό ενισχύει την ε, ιδέα ότι θα ήταν επιθυμητό μέσω άλλων μηχανισμών, ίσως δευτερού πυλώνα, αλλά δεν είμαι ειδικός, να βρούμε τους τρόπους να ευνοήσουμε και άλλα μέτρα που επιτρέπουν τη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου. Κυρίως αναφέρομαι στα μέτρα που βρίσκονται στα αριστερά του γραφήματος και είναι χαμηλού κόστους. Σύνοψη. Η αρχή του πρασινίσματος ε, και του ισοδύναμου βρασινίσματος ε, μπορεί να ευνοήσουν την υιοθέτηση 7 μέτρων μείωσης από τα 26 μέτρα. Αυτό αποτελεί το 23% της συνολικής μείωσης που υπολογίσαμε αν εφαρμόζαμε και τα 26 μέτρα. Δηλαδή, για να έχουμε πιο φιλόδοξους στόχους και να τους πετύχουμε, χρειάζεται ενεργοποίηση και άλλων μηχανισμών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Bardzo Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας. Τώρα μπορεί να ξεκινήσει η συζήτηση και να απαντήσετε. Ο κύριος Άγγιο είναι εδώ πέρα πρώτος ε, στον κατάλογο. Έχετε τον λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν από λίγα χρόνια ε, είχα νιώσει απογοήτευση σε ένα παρόμοιο έργο στο εργαστήριο, με συγχωρείτε και δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αν είναι πραγματικά να αντιμετωπίσουμε τα αέρια θερμοκηπίου, πρέπει να δούμε ποιο είναι το μεγαλύτερο αέριο θερμοκηπίου και είναι ο υδρατμός. και μπορεί να είναι από 65% της ατμόσφαιρας μέχρι καθόλου. Αλλά αν δεν αντιμετωπίσουμε το μεγαλύτερο, δεν έχει νόημα να ασχολούμαστε με το μικρότερο. Όμως κανείς δεν θέλει να μειώσει τους υδρατμούς στον αέρα γιατί είναι τρέλα. Οπότε εάν δεν ασχοληθούμε με αυτό ασχολούμαστε με τα ψηλικά. Διοξίδιο του άνθρακα. 40 μέρη στο εκατομμύριο της ατμόσφαιρας και μία σύγκριση με τους υδρατμούς, αλλά δεν συνειδητοποιεί ο κόσμος πως όσο περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα υπάρχει στην ατμόσφαιρα, τόσο πιο γρήγορα αναπτύσσονται τα φυτά και το αφαιρούν από την ατμόσφαιρα. Δεν έχει νόημα να το μειώνουμε. Έτσι. Και ακούγοντα εδώ πέρα αυτή την παρουσίαση υπάρχει μια ευτυχή σύμπτωση και μια αντίφαση. Η σύμπτωση είναι πως προσπαθώντας να μειώσουμε τι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα ερευνάται τρόπους να μειωθεί η χρήση της ενέργειας. Αυτό είναι θετικό και τουλάχιστον κάτι δικαιολογεί αλλά η αντίφαση είναι φεδρή. Γιατί εδώ πέρα έχουμε το πράσινο λόμπι που μας λέει πως πρέπει να μειώσουμε το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, τη διάβρωση, να έχουμε περισσότερα ψυχανθή, να μειώσουμε τα φυτοφάρμακα και όμως οι επιστήμονες βρήκαν μια λύση. Λέγεται γενετική τροποποίηση. Και το πράσινο λόμπι είναι τελείως κατά. Και ο μόνος λόγος για τον οποίο είναι κατά είναι γιατί μπορεί κάποια εταιρεία μεγάλη να βγάλει κανένα κέρδο. Μα κοιτάξτε, ωραία, ναι. Πράγματι, αν δεν ε, οργώνουμε δεν θα ε, ε, έχουμε διάβρωση. Αλλά βεβαίω εάν δεν έχουμε γενετικά τροποποιημένη τεχνολογία πρέπει να οργώνουμε. Καύσιμα, το ίδιο. Ή γενετικά η τροποποίηση ή περισσότερη χρήση καυσίμων ψυχανθεί. 30 μίλια από το σπίτι μου τους έδωσε ο Bill Gates μία δωρεά για να προσπαθήσουν ε, τις ευεργετικές ιδιότητες των ψυχανθών να την πάνε και στα δημητριακά. Πολύ χρήσιμα πράγματα. Δηλαδή αν είναι να γίνουν όλα τα φυτά έτσι πρέπει να υποστηρίξουν τους επιστήμονες. Τέλος βεβαίως ε, τα ζυζανιοκτώνα δεν σας αρέσουν αλλά αν χρησιμοποιήσουμε αυτή την τεχνολογία μειώνουμε το ποσό ε, των ε, ζυζανιοκτώνων. Κάποια στιγμή πρέπει να αντιμετωπίσετε αυτή την φεδρή αντίφαση. Τώρα, για αυτά τα οποία δεσμεύουν άνθρακα. Θα πρέπει να υπάρχει κάτι το οποίο δημιουργεί εκπομπές, έτσι. Αλλιώς, ξέρω εγώ, ας φυτέψουμε, ξέρω εγώ, συνάπη. Και τι κάνουμε μετά, το κόβουμε, το ξαναπετάμε μέσα και θα ξαναπάει μέσα στο χώμα με άλλη μορφή και ξαναρχίζει ο κύκλος και δεν έχετε κάποιο αποτέλεσμα, έτσι. Τέλος, η μείωση των πρωτεϊνών στο ζωοτροφές. Κοιτάξτε, εγώ ε, εκτρέφω πουλερικά. Χρειάζονται πρωτεΐνες. Οι διατροφολόγοι το ψάχνουν εδώ και 50 χρόνια να βρουν τη σωστή ισορροπία και χοντρικά είναι 1 τρίτο σόγια και 2 τρίτα στάρι. Εάν μειώσουμε τη σόγια όπως προτείνεται, τα πουλερικά μου αντί για 6,5 αυγά της εβδομάδας θα πέσουν στα 6, 5, 4. Οπότε θα χρειάζομαι περισσότερα κοτόπουλα για τα ίδια αυγά, αλλά τα περισσότερα κοτόπουλα κάποια πρωτεΐνη θα δρώνε και αυτά. Οπότε μία ή άλλη. Η ίδια πρωτεΐνη σε περισσότερα πουλωρικά. Δεν έχει νόημα αυτό που λέτε. Ε, ειλικρινά δηλαδή δεν αντιλαμβάνομαι αυτά τα πράγματα. Θέλω μία απάντηση από το πράσινο λόμπι. Αν είστε σοβαροί για αυτά τα οποία λέτε, για τη μείωση της χρήσης ενέργειας, πρέπει να υιοθετήσετε τα γενετικώς τροποποιημένα. <clears throat> Σα ευχαριστούμε. Mm. Είναι μια νέα άποψη για το ζήτημα, θα έλεγα εγώ, ο κύριος Κάπουλα Σάντος τώρα. Και στη συνέχεια ο κύριος Χάουσλινγκ. Πρόεδρε, εγώ δεν θέλω να θέσω ερωτήσεις, γιατί για να το έκανε έπρεπε να έχω διαβάσει και ολόκληρη την έκθεση. Σας άκουσα όμως με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη προσοχή και είδα ότι με πολύ συστηματικό τρόπο μας παρουσιάσατε τις διάφορες εναλλακτικέ λύσεις. Ε, για μας τους πολιτικούς ε, εύκολα είναι να θέσουμε ε, τους στόχους, αλλά το πραγματικό πρόβλημα είναι τα συγκεκριμένα μέτρα που επιτρέπουν υλοποίηση των στόχων πολύ καλή. Η συμβολή σας ε, και ήταν μια σειρά μέτρων και υπομέτρων που μας ε, παρουσιάσατε, άλλα γνωρίζαμε, άλλα όχι. Θα ήθελα, εν πάση περιπτώσει, να σας συγχαρώ για την παρουσίαση. Ήταν πολύ ωφέλιμο το έργο σας. Ε, θα ήθελα παρόλα αυτά να ρωτήσω κάτι που δεν κατάλαβα ακριβώς όταν μιλήσατε για την αποθήκευση της, ε, τη δέσμευση συγγνώμη, του άνθρακα ε, ε, για την αποθήκευση, μάλλον πέρα από δεσμού, για την αποθήκευση του άνθρακα ε, στις διάφορες μορφές του, τι προτείνεται πέρα από τα γνωστά μέτρα. Σας ευχαριστούμε ο κύριος Χάουσλινγκ. Δεν ξέρω αν θα ήθελε και κάποιος άλλος ε, το λόγο μετά, αλλιώς θα είστε ο τελευταίος ομιλητής. Τώρα δεν θα απαντήσω στον κύριο Άγνιο, τα πράγματα είναι αυτεξήγητα. Ήθελα απλά να ρωτήσω, εστιαστήκατε στα μέτρα αναεκμετάλλευση που μπορούν να λάβουν οι αγρότες, αλλά συνολικά νομίζω πρέπει να δούμε και τις ε, εισαγωγές-εξαγωγές. Από το 22 εκατομμύρια εκτάρια ας πούμε που ε, εμείς εισάγουμε, αυτά βρίσκονται, καλλιεργούνται στην Νότια Αμερική και δεν φαίνονται στο δικό μας ισοζύγιο γιατί έχουμε ε, εξαγάγει ουσιαστικά την παραγωγή. Το ίδιο και με τα υπόλοιπα προϊόντα. Ρηπαίνει η Κίνα και εμείς απλά αγοράζουμε τα προϊόντα. Αν είναι δηλαδή να είμαστε έτοιμοι και ειλικρινεί, δεν πρέπει να τα αφήνουμε αυτά εκτός και να λέμε είμαστε πολύ επιτυχημένοι. Δεύτερον, για την παραγωγή αζωτούχων λιπασμάτων που χρειάζεται πάρα πολύ ενέργεια. Φαίνεται αυτό πουθενά. Χαίρομαι που αναφερθήκατε στα ζωτούχα και το αναγνωρίσατε, αλλά έχω την αίσθηση πως ε, οι εκπομπές ε, αυτού του αερίου ε, είναι κάτι το οποίο Βεβαίω δεν λαμβάνεται πολύ υπόψη. Και τέλος όλοι ομόφωνα είπαμε πως ε, θα ήταν ε, μία απάντηση για την ε, επεξεργασία του εδάφους με κάποιο τρόπο ο οποίο το διατηρεί. Αλλά μακροπρόθεσμα νομίζω έτσι εκπέμπεται περισσότερο άζωτο. Δεν νομίζω να λύνουμε έτσι το, το πρόβλημα. Το δείχνουν όλες οι μελέτες πως μετά χρειαζόμαστε περισσότερα ζυζανιοκτώνα Δηλαδή χωρίς Roundup δεν γίνεται, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά κατά κανόνα γίνεται όπως είπαμε η επεξεργασία μέσω της χρήσης συζανιοκτώνων που σκοτώνουν τα πάντα. Δηλαδή φαίνεται ότι κάνουμε κάτι αλλά μακροπρόθεσμα δεν είναι καμία πανάκια δεν ξέρω, μπορεί να τα δηλώσουμε ως περιβαλλοντικά μέτρα. Έτσι, γιατί τελικά πρόκειται για περισσότερη χρήση χημικών προϊόντων. E, Σας ευχαριστώ κύριο Ντες και μετά οι ομιλητές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ αυτά τα οποία μας είπατε. Δεν ξέρω αν έμαθα α, κάποια πράγματα, δεν ξέρω αν αισθάνομαι πιο σοφός. Έχω τέσσερις ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση. Τι γίνεται με τα μέρη του εξωτερικού του ανθρακά ανά εκατομμύριο. Δεύτερον, τι σημαίνει αυτό για τις παγκόσμιες εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα για να δουν συμφέρει. Τρίτον, διαβάζουμε στον τύπο πως είχαμε εκπομπές ρεκόρ διοξιδίου του άνθρακα και κάθε χρόνο έχουμε αύξηση. Γιατί λοιπόν εδώ και 16 χρόνια δεν έχουν ανέβει οι παγκόσμιες θερμοκρασίες. Τέταρτον, γνωρίζω από τα βιβλία της ιστορίας πως στο νότο τουλάχιστον της Γερμανίας παλαιότερα το 1 τρίτο της καλλιεργήσιμης γης το άφηναν χέρσο. Αλλά τη χρονιά που το άφηναν χέρσο το όργωναν 4-5 φορές για να είναι έτοιμο. Παρά το ότι ε, γινόταν ε, και γίνεται αυτό γιατί ε, εξακολουθεί να, εξακολουθούμε να έχουμε περισσότερο κρύο. Δεν νομίζω να οφείλεται αυτό στο όργωμα. Έτσι δεν είναι πολύ λογική η εξήγησή σας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Οι ομιλητές νομίζω μπορούν να κανονίσουν μεταξύ τους ποιος θα απαντήσει πρώτα. Merci. Euh, Ευχαριστώ. Να δώσω μια πρώτη απάντηση ε, που αναφέρεται ταυτόχρονα στην ερώτηση του κυρίου Άγνιου και στην ερώτηση του κυρίου Στην ε, μελέτη που σας παρουσίασα, όπως ε, διευκρίνησα και στην αρχή, εξετάσαμε μέτρα υπό την προϋπόθεση ότι δεν μειώνουν τις αποδόσεις της συγκομιδής. Υπάρχει ένα μικρό ποσοστό ανοχής στη μείωση των αποδόσεων, αλλά είναι αμεληταίο. Διότι δεν επιθυμούσαμε να επικεντρωθούμε σε μέτρα μείωσης των αποδόσεων, εφόσον έτσι θα μεταφέραμε το πρόβλημα σε άλλες υπήρους. Μπορούμε εν ίδια να πούμε ότι για να μειώσουμε δραστικά τις επιπτώσεις των αερίων θερμοκηπίου μια ιδανική λίστα ήταν να ε, σταματήσουμε τη γεωργική δραστηριότητα εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να εισάγουμε όλα τα προϊόντα. Αστειεύομαι, δεν είναι φυσικά αυτή η λύση που προκρίναμε στο Ινστιτούτο μας, στο Ίνερα. Οριακή λοιπόν είναι η μείωση ε, στις αποδόσεις όλων των μέτρων που εξετάσαμε στα πλαίσια της μελέτης μας. Για την ε, αύξηση της αποθήκευσης ε, άνθρακα στις γεωρικές γης είναι ξαναλέω ένα εργαλείο, ένας τρόπος, ένας μοχλός για να επιτύχουμε ένα αποτέλεσμα. Ποιο είναι το αποτέλεσμα, η γεωργία με θετικό τρόπο να συμβάλλει στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Δηλαδή η γεωργία πλέον δεν εκλαμβάνεται μόνο ως παραγωγός αερίων, αλλά ε, συμβάλλει στην καταπολέμηση του φαινομένου ε, του θερμοκηπίου. Και άρα προσφέρει μια διαφορετική υπηρεσία στην κοινωνία. Εξετάσαμε λοιπόν τους τρόπους αποθήκευσης του άνθρακα είτε αυξάνοντας ε, τις, ε, τους τρόπους εισόδου. Ξέρετε ότι με τη φωτοσύνθεση τα φυτά δεσμεύουν ε, τον άνθρακα και επιστρέφει στη γη, στο έδαφος ο άνθρακας, ένα μέρος του τουλάχιστον, ε, αποθηκεύεται με μόνιμο τρόπο. λοιπόν, οι τεχνικές ε, φυτοκάλυψης, όλες οι τεχνικές φυτοκάλυψης, ε, ε, αποσκοπούν ακριβώς στην μείωση της εισόδου άνθρακα στο έδαφος. Στη συνέχεια, ελάττωση της ορυκτοποίησης το άνθρακα και επιστροφή του ε, στην ατμόσφαιρα. Ε, αυτό γίνεται με επιβράδυνση ε, της διαδικασίας. Δηλαδή επιβραδύνουμε την επιστροφή στην ατμόσφαιρα και παρατείνουμε την περίοδο την οποία παραμένει μέσα στο έδαφος ο άνθρακας. Μέσα στην βιομάζα λοιπόν έχουμε την αγροδασοκομεία, Ε, το steady state, ε, η ε, πυκνή δεντροφύτευση παραδείγματος χάρη είναι ένας άλλος τρόπος όταν διαρκώς αλλάζεται την δεντροφύτευση τότε μειώνονται τα αποτελέσματα. Όταν είναι steady state, δηλαδή διατηρείται η δεντροφύτευση ως έχει, τότε έχουμε τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα. Συνεχίζω συνάδελφος. Εγώ θα συμπληρώσω σε σχέση με τα πλεονεκτήματα που μπορεί να υπάρχουν και τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις από τη μείωση των εκπομπών. Τα τελευταία τρία χρόνια συνεργαστήκαμε πάνω από 120 γεωργούς και η εμπειρία μας είναι ότι αν εργαζόμαστε σε κοινά σχέδια δράσης στα πλαίσια μέτρων που εξηγήθηκαν εδώ δεν είναι τίποτα παραπάνω παρά από τη βελτίωση της γνώσης που έχει ο Γιώργος για την εκμετάλλευση και είναι εκπληκτικό να δούμε πώς το να συνοδεύουμε τους Γιωργούς στην εφαρμογή αυτών των μέτρων τελικά οδηγεί σε καλύτερη γνώση του Γιωργού για τη λειτουργία της εκμεταλλευσής του, σε καλύτερη γνώση των περιορισμών και των ευκαιριών. Επομένω, ε, καλύτερη θέση του Γιωργού απέναντι στο μέλλον. Και όπως είπε και ο κύριος Πελέρα, τα μέτρα στα οποία επικεντρωθήκαμε κυρίως είναι πράγματι τα μέτρα που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα των γεωργών. Εργαστήκαμε με 120 150 συγγνώμη λέει τώρα μιλητές, ε, γεωργούς για τρία χρόνια και τα μέτρα αυτά εκτελέστηκαν ουσίως και το να εφαρμόζει εκούσια ένα γεωργό τα μέτρα αυτά είναι επειδή έχει κάποιο όφελο. Δεν θα τα εφαρμόσει αν δεν ωφελεί την εκμεταλλευσή του αυτό. Επίση, υπάρχουν μια σειρά πλεονεκτημάτων και συνεργειών που δεν μπορούμε να αρνηθούμε και επιπρόσθετα θα μπορούσαν πολύ καλά να ενταχθούν στη σημερινή αλλά και στη μελλοντική δομή της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής. Εμείς ε, κάναμε αυτή την ε, άσκηση για να εργαστούμε όχι μόνο στα μέτρα του περσινή αλλά να δούμε και ποιο είναι το σύνολο των μέτρων που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο δεύτερο πυλώνα ή μάλιστα και ενισχύοντας τη σημερινή αιρεσιμότητα ή πολλαπλή συμμόρφωση. Υπάρχουν πολύ σημαντικές συνέργειες που επιτρέπουν ή που μας, ε, μας επιτρέπουν να αξιολογήσουμε τα μέτρα αυτά. Και για να απαντήσω στην ερώτηση του κυρίου Κάπουλα Σάντος, σε ό,τι αφορά το διοξείδιο του άνθρακα, πέρα από την αποθήκευση του άνθρακα στο έδαφος, τα συμπεράσματά μας ε, ήταν ότι αν και τα μέτρα που επικεντρώνονται στην ενέργεια είναι αυτά τα οποία θα έχουν το μεγαλύτερο ε, αντίκτυπο στο επίπεδο εργοσία, ε, επίπεδο είναι και αυτά που υποδέχονται καλύτερα οι γεωργοί, γιατί ουσιαστικά συσχετίζουν ε, την εξοικονόμηση σε επίπεδο ενέργειας, ε, την εξοικονόμηση σε επίπεδο πόρων και την βελτίωση της μείωσης των εκπομπών. Και αν θέλουμε να μιλάμε για την μείωση των εκπομπών σε επίπεδο εκμετάλλευσης, η γεωργοί είναι αυτή που θα θέσουν σε εφαρμογή αυτά τα μέτρα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε κατά νου μέτρα που θα ευνοούν και το δυναμικό, αλλά και μέτρα που θα θεωρήσει ο Γιωργός εύκολα, χρήσιμα και επομένως μιλάμε όχι μόνο για τεχνικές πτυχές, αλλά και για οικολογικές, ψυχολογικές διορθανομιλητές. Και σε σχέση με τις συγκεντρώσεις διεξουδίου του άνθρακα, όταν εργαζόμαστε με τους γεωργούς ένα ε, περίοδο, δεν ξέρουμε ποια είναι η συγκέντρωση διεξουδίου του ανθρακά στην ατμόσφαιρα. Δεν έχει σημασία για μας, αλλά εμεί ξέρουμε ότι ολοκληρώνει συγκεκριμένη περίοδος και έχουν εκτελεστεί ορισμένα μέτρα. Ο γεωργός αυτός έχει αποκτήσει οικονομικό πλεονέκτημα, καλύτερη απόδοση, έχει εξοικονομήσει χρόνο και άλλα ωφέλη. Έτσι λοιπόν, αν ε, η μείωση των εκπομπών ε, ουσιαστικά συνδέεται με την αύξηση και των εσόδων του γεωργού, τότε αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Να απαντήσω στο σχόλιο του κυρίου Χόσλινγκ. κάτι φορά ε, του υπολογισμού των ε, εκπομπών, ναι, λαμβάνουμε υπόψη ότι ε, μπορούν να, να συνεισφέρουμε στο δυναμικό της μείωσης των εκπομπών που προτείνεται. Και σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα, εμείς ε, βλέπουμε ποιες είναι οι πηγές των εκπομπών ε, και τις εκπομπές ανάντι. Και δεύτερο συμπληρωματικό στοιχείο σε ό,τι αφορά τη γεωργία συντήρησης πρόκειται για ένα από τα μέτρα που προτείνουμε και θα μπορούσαμε να έχουμε μια αλλαγή σε ό,τι αφορά τα παρασιτοκτόνα. Γι' αυτό έχουμε επιμείνει στην έκθεση και εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει ουσιαστικά μια ε, σύνθεση μέτρων από το Γεωργό για να μειώσει τελικά και τη χρήση των παρασιτοκτόνων. Ευχαριστώ πολύ. Φτάνουμε τώρα στο τέλος αυτής της συζήτησης. Και φυσικά όλα όσα υπόθηκαν εδώ συνδέονται και με οικονομικά ζητήματα. Και φυσικά υπάρχουν και προσδοκίες από τον Ευρωπαίο Φορολογούμενο και για και για το γεωργικό τομέα και όταν μιλάμε για την γεωργική πολιτική πρέπει να δούμε ποια είναι τα καλύτερα μέσα για το πρασίνισμα. Και να προσπαθήσουμε εμείς ε, και ως Κοινοβούλιο αλλά και Κομισιόν να καταλήξουμε σε ένα κοινό συμβασμό. Αγαπητοί συνάδελφοι, και πάλι σας ευχαριστώ όλους. Ευχαριστούμε και το τμήμα πολιτικής για την οργάνωση αυτού του τόσο ενδιαφέροντος σεμιναρίου και φτάνουμε τώρα στο τέλος των εργασιών μας για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε στις 27 Ιανουαρίου. Καλό βράδυ σε άλλους και τα ξαναλέμε την επόμενη φορά.